Good afternoon to all of you. Καλησπέρα σας. Ελπίζω να φάγατε καλά το μεσημέρι. Εγώ έφαγα πάντως πολύ καλά. Και τώρα θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Μακρά η σημερινή ημέρα, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα. Εξαιρετική και η πρωινή ακρόαση. Μας έδωσε πολύ τροφή για σκέψη και συζήτηση για τις επόμενες ημέρες. Να σα αναφέρω ποιε είναι οι ανακοινώσεις ε, του πρόεδρου σχετικά με τι αποφάσει των συντονιστών. Σχέδιο ημερήσια διάταξη για 14 Ιουλίου. Εγκρίναμε με τις εξή αλλαγέ στη ημερήσια διάταξη. Η κυρία Μακίνες ε, θα προσκληθεί στην Επιτροπή μα ε, ω διαμεσολαβήτρια για τα δικαιώματα των παιδιών. Συμμετείχε σε μια συνεδρία στο Λονδίνο για τα θέματα που αφορούν τα παιδιά και θα μα αναφέρει ποια ήταν τα πορίσματα αυτής της συνάντησης, ε, αιτήματα για τη μέση διάταξη του Ιουλίου, θα περιληφθούν τα αιτήματα των πολιτικών ομάδων και στη μέση διάταξη του Σεπτεμβρίου. Δεν με ακούτε? Σας ακούω, αλλά διαφωνώ, λέει κύριε Άουκεν. Για τους συντονιστές, μπορώ να σας πω πρώτα. Ναι, μου είπαν όμως τι έγινε χθε και διαμαρτύρομαι. Πρόεδρος, θα σας δώσω το λόγο όμως αφού ολοκληρώσω. Λοιπόν, για την σε του σε τέσσερι αναφορές για τα άτομα με αναπηρία. Το πρώτο, ε, μάλλον ένα θέμα για την αστική ανάπτυξη στην περιοχή ΒΑΡ. Ένα για την κατασκευή ενός χώρου μην τάφης απορρίμματων στη Βουλγαρία. Ίσως συζητηθεί αργότερα. Και ξέρω ότι αυτό είναι το θέμα που θέλετε εσείς να συζητήσουμε. Μα περιμένετε μισό λεπτό. αναφέρουν έχει ε, παράσχει νέες πληροφορίες. Τις έχει λάβει και η Κομισιόν τις πληροφορίες αυτές. Η Κομισιόν ξεκαθάρισε στη γραμματεία ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο για το θέμα αυτό. Αν θέλετε οι πράσινοι να το επαναφέρετε στην σχεδιάταξη το ζήτημα, πρέπει να μας το αιτιολογήσετε πλήρως. Ποια είναι αυτά τα νέα ευρήματα που ενδεχομένω έχετε και τα οποία επαρκούν ώστε να ε, με σχέδιο στο θέμα. Δεύτερον, έγκριση προφορική ερώτηση για την νομοθεσία περί στεγαστικών δανείων και κάποιων ε, άλλων ε, χρηματοπιστωτικών εργαλείων κινδύνου. Αποφασίσαμε γι' αυτό. δύο φορούν στην Ισπανία. Να έχουμε μία προφορική ερώτηση και για τα δύο ζητήματα. και επεξεργάζεται το σχετικό κείμενο γραμματεία. Θα αποτελέσει δε αυτό το κείμενο τη βάση για την προφορική ερώτηση για να μπορέσουμε να την εγκρίνουμε τον Ιούλιο. Έχουμε προθεσμία κατάθεση τροπολογιών που λύγει την Τρίτη στις 30 ε, του μήνα, επόμενη Τρίτη δηλαδή, σε 6 το απόγευμα. Άρα έχετε μια εβδομάδα για να εργαστείτε για αυτό το ζήτημα. 15 προτάσεις το πολύ. Δεν ελήφθη απόφαση για πιθανό σχέδιο ψηφίσματο που ολοκληρώνει την σχετική συζήτηση. Σε ό,τι αφορά τι προσβαλόμενε συστάσει οι συμβαστικές λύσεις που πρότεινε η πρόεδρος σας έγιναν δεκτές χωρίς καμία εξαίρεση και αποφασίστηκε να ζητηθεί νομική γνωμάτευση για το παραδεκτόν ή μη της ε, προσβαλόμενης συστάσεως ε, για αναφορές που αφορούν το Jugendamt στη Γερμανία. Αυτά ήταν. Ε, εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αποφάσεις αυτές για εκθέσει και γνωμοδοτήσει ε, συντονίτρια και καμπεθών από τη ε, ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών αργότερα σήμερα. Θα σα ενημερώσει για την απόφαση τη ομάδα τη κατά πόσο θα αναλάβει την έκθεση ή όχι για την ε, ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων τη Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτρια για το 2014. Είναι έξω και περιμένει να μπει στην αίθουσα για να μα αναφέρει τα σχετικά σημεία 5 με 12 επειδή δεν υπήρχε διερμηνία. γραπτή διαδικασία θα ακολουθηθεί για τα θέματα αυτά. Και τώρα έχω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Την χάνει να είμαι η εισηγήτρια στην ε, Λίμπε και τη Δευτέρα το απόγευμα συνδράζουν συντονιστές ε, στο Στρασβούργο για δύο-δυόμιση ώρες κάθε φορά. Στη δική μας την Επιτροπή για τους συντονιστές προβλέπεται συνεδρίαση διάρκειας μιας ώρας. Και επειδή μιλάει ο κόσμο εδώ στην Επιτροπή, και καλό είναι αυτό βέβαια, καθυστερεί να αρχίσει να συντονιστών πιο πολλέ φορέ και άρα ούτε αυτή την ώρα δεν την έχουμε στη διάθεσή μα. Επομένω είναι αδύνατο να ασχοληθούμε με όλα τα θέματα μέσα σε μια ώρα. Αποφάσισα λοιπόν να προσπαθήσουμε να αναδιοργανώσουμε τη συνέντευξη των συντονιστών ώστε να επιτρέψουμε να γίνεται μια πλήρη συζήτηση, να συζητούνται τα θέματα και όχι απλά να τα αντιμετωπίσουμε στο πόδι. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι η Επιτροπή μας πρέπει να εργάζεται στο ίδιο επίπεδο, ε, σε ισότιμο επίπεδο με άλλες επιτροπές. Στη Γιούρη και Λίμπε που έχω υπάρξει συντονίστρια πάντοτε είχαμε αρκετό χρόνο για να μπορούμε να εργαστούμε αποτελεσματικά. Οι πράσινοι πάντως καίγονται να πάρουν το λόγο. Γι' αυτό το λόγο σας καταλαβαίνω και συμφωνώ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι όταν έχουμε τόσο δύσκολους και στενούς, στενά χρονικά περιθώρια να μπορώ να τα φέρω σε πέρα όλα τα θέματα. Αυτά λοιπόν για την συνδρίωση των ανταγωνιστών. Κύριε Τέρη Κάμπρας, έχετε τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ. Είπατε σωστά το όνομά μου για μια φορά. Σας ευχαριστώ. Το μάθατε. Είναι δύσκολο το όνομά μου, το ξέρω. Σας ε, παραπέμπω στη σχετική συνεδρία των συντονιστών που είμαστε όλοι εξαντλημένοι, κουρασμένοι και ίσως και αυτό ήταν η αιτία κάποιων παρανοήσεων ή παρερμηνιών. Μας είπατε, μας είπατε στην ομάδα των Πρασίνων και της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας ότι είμαστε πολύ ωραίοι. Και σας είπα ναι, το ξέρω ότι είμαστε πολύ ωραίοι αλλά το είπα αφού είχατε δεχθεί ότι το σημείο μας ε, σε ό,τι αφορά το πιλωτικό πρόγραμμα να συζητηθεί τι τον Ιούλιο. Και έχω μάρτυρες εντός της αιθούσης. Δεχτήκατε να συζητηθεί τον Ιούλιο. Μετά αποφασίσατε να γίνει το Σεπτέμβρη η συζήτηση. Και σοκαρίστηκα ξεπλάγει, διότι η πρώτη σας απόφαση, δική σας απόφαση ήταν για τον Ιούλιο. Γι' αυτό και έλεγα εγώ ότι είμαστε όλοι ωραίοι και εσείς είστε ωραίοι και όλα είναι ωραία και καλά. Για το δεύτερο ζήτημα, το βουλγαρικό, το δέχομαι. Αποφασίσατε ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα είπαμε γιατί δεν έχουμε έγγραφα για να δείξουμε που να τεκμηριώνουν τις ε, δικές μας προτάσεις. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη και αυτό συνδέεται με την ερώτηση που έχει γραφεί. Το ενδεχόμενο ψηφίσματος. Από τί είδα εδώ, τέσσερις πολιτικές ομάδες ήταν υπέρ της κατάθεσης ψηφίσματος. Μία ομάδα δεν ήταν υπέρ, αλλά δεν τέθησε ψηφοφορία το θέμα και εσείς αποφασίσατε να μην έχουμε ψήφισμα. Γι' αυτό λοιπόν και στις δύο περιπτώσεις, το αφορά το πλειοτικό και το δεύτερο για ε, το ψήφισμα πρέπει να διαφωνήσω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο καλός είμαι και θα δεχθώ αυτά που λέτε τελικά. Έχω όμως το δικαίωμα και το καθήκον να πω τι συνέβη ακριβώς και να εκφράσω τη διαφωνία. Πρόεδρος. Απολύτως έχετε κάθε δικαίωμα να πάρετε το λόγο και να διαφωνήσετε. Και εγώ συμφωνώ. Για το ΒΑΡ ε, αφισβητήθηκε από τις άλλες ομάδες, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να το συμπεριλάβουμε στην ημερήσια διάταξη και σε ό,τι αφορά την ε, δεύτερη παρατήρησή σας για το αν θα υπάρξει ψήφισμα ή όχι, νομίζω, δεδομένης της εμπειρίας που έχω, Έπρεπε να το συζητήσουμε ανοιχτά. Είτε θα είχαμε δύο προφορικές ερωτήσεις, αλλά αυτό που είπα εγώ είναι ούτε για μια στιγμή δεν θα μπορούσε η διάσκεψη των Πρόεδρων να σκεφτούμε ότι θα εγκρίνει δύο προφορικές ερωτήσεις. Γι' αυτό λοιπόν ε, για την πρόταση ψηφίσματος είπαμε ότι μία ομάδα μπορεί να υποβάλει πρόταση ψηφίσματος. Αυτό υπόθηκε ξεκάθαρα και κατά δεύτερον είπα ότι έχω σοβαρούς ενδιασμούς για το κατά πόσον θα περάσει από τη διάσκεψη των Προέδρων και προφορική ερώτηση και ψήφισμα. Εάν όμως υποβάλλουμε πρόταση για ψήφισμα, είπα ξεκάθαρα ότι θεωρώ ότι ο καλύτερος τρόπος να το χειριστούμε θα ήταν να γίνει αυτό με ανάλογη ενέργεια και εξέταση του θέματος από Επιτροπή με νομοθετική αρμοδιότητα. Θα έπρεπε να στραφούμε και προς αυτούς. Όμως κανείς δεν ήθελε να το κάνω αυτό. Ήμουν έτοιμη να στείλω επιστολή προς την Επιτροπή ΕΚΟΝ και να ζητήσω να γίνει βάση του άρθρου 54-55. Αλλά αποφασίσαμε στην Επιτροπή και εδώ είναι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, μπορούν να το επιβεβαιώσουν και οι συνάδελφοι της Γραμματείας, αποφασίσαμε να υποβάλουμε προφορική ερώτηση και το ψήφισμα να το αφήσουμε για κατοπινό στάδιο. Όμως δεν ήταν αυτή η δική μας η θέση και δεν ψηφίστηκε. Ε, λοιπόν έπρεπε να έχουμε το δικαίωμα να εκφράσουμε τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν. Νομίζω η άποψη της πλειοψηφίας ήταν υπέρ του ψηφίσματος. Με συγχωρείτε, δεν μπόρεσα να είμαι παρούσα χθε, αλλά άκουσα όσο είπε ο Ζανμαρή και πρέπει να πω ότι κλείσωμε κάπως στι ομάδες. Ε, δεν συνεννόμαστε έτσι μεταξύ μα. Εγώ τα πληροφορήθηκα και ακούω από τον Ζωζέ Μαρία, από τον Χωσέ Μαρία, ότι για την περίπτωση της Βουλγαρίας, εγώ πήγα σε αυτή την αποστολή για την ε, εξέβεση στοιχείων στην Βουλγαρία και πρέπει να πω ότι έχει πάρει διαστάσεις στο θέμα αποφασίσαμε το θέμα να μην κλείσει, να εξεταστεί περαιτέρω. Και πραγματικά μας φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση το γεγονός να έχει ληφθεί τέτοια απόφαση και να έχουν κατακλειστεί οι άνθρωποι στη χωματερία αυτή από επικίνδυνα απόβλητα. Δεν είσαστε εκεί. Εγώ ήμουν. Ήμουν και είδα τι συμβαίνει δεν μπορούμε απλώς επειδή σε εσά δεν σας αρέσει ή γιατί εσείς πιστεύετε ότι είμαστε μικρότερη σημασία ομάδα να μην προχωρήσει. Δεν μ' αρέσει αυτός ο τρόπος εργασίας. Αποφασίσαμε να παραμείνει ανοιχτό το θέμα. Αποφασίσαμε να το εξετάσουμε περαιτέρω και εσείς αποφασίσατε το αντίθετο. Πρέπει να διαμαρτυρηθώ και γι' αυτό λοιπόν. Exactly. Ακριβώς. Αυτό προέκυψε λόγω του μπαλαγιάζ. Έτσι είναι, αλλά εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη γραμματεία μας και εφόσον συνεννοήθηκαν με την Επιτροπή ότι δεν υπάρχει καμία νέα ουσία, αποφασίσαμε κι εμείς και βάσει των κανόνων ότι αν δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ή πληροφορίες που να αλλάξουν την όλη εξέταση του ζητήματος, τη θέση μας προς το ζήτημα, θα πρέπει η ομάδα να, έχει, να δώσει πλήρη τεκμηρίωση για να συμπεριληφθεί και πάλι στην ημερήσια διαταξή. Κοιτάξτε, σε αυτή τη φάση έχω την αίσθηση ότι μας πιέζει και ο χρόνος. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Μεσολαβήτρια να μας ε, περιμένει. Θέλετε να συνεχίσουμε από αυτού ή όχι. Κοιτάξτε, πραγματικά είναι πολύ δυσάρεστο, αλλά έχω την αίσθηση και το έχω δει και εγώ η ίδια, ότι εάν δεν σας αρέσει μια απόφαση ή δεν σας αρέσει αυτό που σας ε, λέει η γραμματεία, περνάτε απευθείας στο επόμενο θέμα. Ακούστε με πρόεδρε, ε, μπορείτε να αλλάξετε την ε, όλη μας θέση. Δεν αισθάνομαστε ασφάλεια με αυτόν τον τρόπο διεξαγωγής της όλης συζήτησης. Ξέρουμε ότι δεν σας αρέσει να μείνει έτσι το θέμα της Βουλγαρίας, αλλά εμείς έχουμε ασχοληθεί πολύ σοβαρά με αυτό το θέμα. Δεν μπορείτε να μας ε, αναγκάζετε να μην κάνουμε τίποτα για αυτό το θέμα. Υπάρχουν αναφορές σχετικά, πρόεδρος. Εντάξει, προσωπικός, θα δω ποια είναι αυτά τα νέα στοιχεία, τι ε, νέες πληροφορίες έχουν προσταθεί στις παλιές και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Να δώσω το λόγο στον Πίτερ και μετά στον Γιάρεκ. Να πω κάτι για τον κανονισμό. Συγγνώμη, διακόπτη Διακόπτεται ο μίλητης. Κάναμε την συνάντηση των συντονιστών και έγιναν διάφορες αποφάσεις λήφθησαν. Δυστυχώς και πάλι μιλούν πάνω στον ομιλητή υπόλοιπη. Προσπαθήσαμε να βρούμε ένα χρόνο... Διακόπτεται το μικρόφωνο, το ομιλητή. Είναι πολλά τα μικρόφωνα που είναι ανοιχτά, οπότε έτσι δεν μπορεί να γίνει διερμηνία. Δεν σας είδα να ζητάτε το λόγο. Από την αρχή, Πρόεδρε. Okay. Peter, would you mind giving the floor to, to Mrs. Valina? Πέτερ, αν δεν έχει αντίρρηση, να δώσουμε το λόγο στην κυρία Βαλίνα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μου παραχωρεί το λόγο ο κύριο Γιάρ, βέβαια, γιατί είχα ζητήσει από την αρχή το λόγο. Τέλο πάντων, θέλω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την ε, παρέμβαση των συμπαθέστατων πρασίνων. Δεν ξέρω αν ε, στην ΚΟΥ είμαστε τόσο συμπαθητικοί και τόσο ωραίοι όσοι πράσινοι, αλλά χθε και σήμερα, τέλο πάντων, μιλήσαμε για τη σημασία που έχουν οι αναφορέ, ε, για τη συμμετοχή των πολιτών, ότι θα πρέπει τα θεσμικά οργανά να είναι ανοιχτά προ του πολίτε κτλ. Και τι κάνουμε εδώ, το αντίθετο. Ποτέ δεν έχουμε χρόνο να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να ολοκληρώσουμε ε, την μέσια διάταξη τη συνεδρίασης των συντονιστών, να τρέχουμε συνέχεια, βιαζόμαστε, πηδάμε το ένα σημείο της μέσης διάταξης στο άλλο και χθε πράγματι Υπήρχαν τέσσερι πολιτικέ ομάδε που θέλαμε και προφορική ερώτηση και ψήφισμα. Πράγματι, είχαμε στήσει αρχικά δύο προφορικέ ερωτήσει. Δεχθήκαμε να γίνει μία προφορική ερώτηση, το είπαμε και από την αρχή τη συνεδρίαση. Τέσσερι όμω πολιτικέ ομάδε θέλαμε και ψήφισμα. Και δεν μα επιτράπει ούτε να ψηφίσουμε ούτε να εκφραστούμε. Ότι να πούμε και τέσσερι πολιτικέ ομάδε τι θέλουμε. Αυτό δεν είναι δημοκρατική διαδικασία στις συνεδριάς. μετά μένουμε χωρίς διερμηνείς, ε, είμαστε τελευταίοι στην ουρά για διερμηνείς και για όλα. Δεν μπορεί να λέμε σε μια μερίδα σήμερα το πρωί πόσο σημαντική είναι η Επιτροπή μας και πόσο σημαντικό είναι το δικαίωμα αναφοράς και έπειτα καθημερινά να αποδεικνύουμε το αντίθετο. Σας διαβεβαιώ ότι θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε περισσότερο χρόνο για τους συντονιστές. Μια καλύτερη χρονοθυρίδα Συμφωνώ απολύτω μαζί σας και πραγματικά στενοχωριέμαι ίσως και περισσότερο από εσά την ίδια. Ε, δεν είναι ευχάριστο να έχουμε συνεδριάσεις και πίεση χρόνου για να μην προλαβαίνουμε την ημερήσια διάταξη και να μην προλαβαίνουν όλοι να τοποθετηθούν. Γιάρεκ. Όχι, όχι, με συγχωρεί, Και μετά ο Γιάρεκ. Για τον κανονισμό ήθελα να πω κάτι γιατί ανησυχώ από την άλλη. Μία έχουμε τους ε, προέδρους των επιτροπών ε, που δεν έχουν αρκετό χρόνο για τους συντονιστές λόγω της παράτασης των ε, συνεδριάσεων. Ε, πολλές φορές αρχίζουμε με καθυστέρηση, δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Ένας κατηγορεί τον άλλον. Αυτό που δεν γίνεται όμως, αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να ξεκινήσει και πάλι η συνάντηση των συντονιστών γιατί δεν έχουμε σήμερα τέτοια συνάντηση. Γιατί είμαστε κατά του ψηφίσματος ας πούμε. Γιατί θέλαμε να μην υπάρχει ε, ψήφισμα. Αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Τώρα έχει τελειώσει αυτή η συζήτηση. Ίσως να ε, σβήσουμε το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης ε, για να γίνει αυτό μετά. Υπάρχει ε, η διαδικασία ε, που επαναλαμβάνεται και θα μπορούσαμε να με την επαναλάβουμε. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Κάνουμε τη συνάντηση των συντονιστών, γίνονται οι αποφάσει, λαμβάνονται οι αποφάσεις και μετά γίνονται όλα τρεις και δύο φορές και τρεις γιατί δεν συμφωνούμε. Ε, καλό θα είναι λοιπόν αυτά να τα ξεκαθαρίσουμε οι πράσινοι κάνουν το ένα, οι άλλοι κάνουν το άλλο. Ο πρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να διαπιστώνει κάθε φορά ποια είναι η κατάσταση, να γίνονται όλα αργά, να το κάνουμε στην συνάντηση των συντονιστών κάθε φορά να μπορούμε να εξετάσουμε όλα τα σημεία όπως έπρεπε και όταν κάτι ε, βγαίνει να, να μπορούμε κάποια στιγμή να το συζητάμε, να μην πάνε όλα μέσω γραπτής διαδικασίας. I agree with Peter. We should move Εγώ συμφωνώ με τον Πίτερ, θα πρέπει να προχωρήσουμε από το σημείο και πραγματικά είναι κρίμα που κάνετε την ατμόσφαιρα τη συνεδρίαση. Οι περισσότεροι συντονιστέ που ήταν χθε στη συνεδρίαση σήμερα δεν βρίσκονται εδώ. Είναι αδύνατο λοιπόν να αντικρούσουμε τα επιχειρήματά σα. Α προχωρήσουμε τέλο πάντων στην επόμενη συνεδρία των συντονιστών το θέμα αυτό και α συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη. Διότι σε αυτή τη φάση δεν έχει νόημα να συνεχίζεται αυτή η συζήτηση. Ε, πρόεδρος, ε, έτσι είναι. Θα τα δούμε τα θέματα αυτά με γραπτή διαδικασία και θα προσπαθήσω να προβλέψω καλύτερες χρονοθυρίδες στο μέλλον. Θα ήθελα τώρα να γυρίσετε τη σελίδα και να στρέψετε και το νου σας στους προκεκλημένους που έχουμε στην αίθουσα. Βλέπετε ότι όλα γίνονται διαφανώς εδώ. Είναι η Επιτροπή μας μια από τις πλέον δραστήριες ε, στο Κοινοβούλιο. Υπάρχουν ε, φωνές, κομμή, αλλά τελικά το πνεύμα συνεργασίας νομίζω ότι είναι αγαστό και τα αποτελέσματά μας θετικά. Ε, θα δούμε λοιπόν, ε, ε, έχουμε μαζί μας προκεκλημένους από την Εθνοσυνέλευση της Ουαλίας και με τον πρόεδρο τον κύριο Πάουελ να ηγείται. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Αναφορών μας. Και είναι μεγάλη μας χαρά που σας είχαμε εδώ από το πρωί για την ακρόαση που είχαμε. Θα θέλαμε να σας ακούσουμε για μια ομιλία, παρέμβαση, κάτι τέτοιο, αλλά έχουμε εδώ και την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, που εντελώς κατά τύχη είναι και Ιρλανδή. Ε, περιμένει απ' έξω. Και εκείνη την πιέζει ο χρόνος. Γιατί λοιπόν να μην έχουμε αυτή την ωραία ανταλλαγή φιλοπρονήσεων μετά, εάν συμφωνείτε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν, καλώς ήρθατε, χαιρόμαστε που είστε σήμερα εδώ και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί σας και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα μπορούσε κανείς να φέρει μέσα την Έμιλη. Λοιπόν, καλώς ήρθατε κυρία Οράιλη στην Επιτροπή Αναφορών. Αυτή είναι εδώ η έκθεση από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Είναι η πρώτη της ε, έκθεση πεπραγμένων για το πρώτο έτος της, της, θητεία της, της μετά την ε, επανεκλογή της ε, τον Δεκέμβρη πέρυσι. Συγχαρητήρια λοιπόν η εικόνα στο εξώφυλλο είναι ενδιαφέρουσα. Ε, πραγματικά αξίζει να την ε, δούμε και να τη σκεφτούμε. Στην έκθεση εκφράζει την ικανοποίησή της για τα αποτελέσματα της έρευνας όσον αφορά στην διαφάνεια της ε, TTIP, των ε, διαπραγματεύσεων δηλαδή για τη Διατλαντική Συμφωνία και για την κοινή προσπάθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αύξηση της διαφάνειας ε, στις ομάδες πίεσης. Έχουν γίνει διάφορε έρευνε για αυτό το θέμα ε, όσον αφορά ε, τη σύνθεση και τη διαφάνεια των ομάδων εμπειρογνωμόνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το φαινόμενο τη μεταπίδηση από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα. Έχει γίνει μία έκθεση από την Επιτροπή μας για τις δραστηριότητές σας το 2014, όμως τώρα σας δίνω το λόγο για να μας κάνετε ε, κάποια ξενάγηση, ας πούμε, σε αυτήν την ετήσια έκθεση πεπραγμένων. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ και εγώ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Είναι χαρά μου που βρίσκαμε εδώ και ιδιαίτερα επειδή όπως είπατε παρουσιάζω την πρώτη μου έκθεση πεπραγμένων η οποία εκπροσωπεί το πρώτο έτος ε, εργασίας. Να σας πω ποια είναι τα βασικά σημεία της έκθεσης. Όσοι με έχετε γνωρίσει ήδη θα ξέρετε ότι ένα από τα πράγματα που κάνω στο γραφείο μου είναι να επικεντρώνομαι ειδικότερα στις δικές μου πρωτοβουλίες όσον αφορά τις ε, ατομικές καταγγελίες αλλά ταυτόχρονα θέλω να ξεριζώσω αν θέλετε ζητήματα συστημικής ε, κακοδιαχείρισης και σε αυτή την παρουσίαση θα σας δείξω πολλές από αυτές τις υποθέσεις ε, τις οποίες αντιμετώπισα το τελευταίο έτος. Εδώ λοιπόν έχουμε μια επισκόπηση του 2014, τα βασικά γεγονότα. Για παράδειγμα, τον Αύγουστο είχαμε την ε, ε, ιδίας πρωτοβουλίας έρευνα για τη διαφάνεια στη Συμφωνία TTIP Επίσης, ε, η καταγγελία στο Σεπτέμβρη, το θέμα της μεταπίδησης από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, το revolving doors όπως ονομάζεται, ας πούμε η άνθρωποι που φεύγουν από ψηλά αξιώματα στο δημόσιο και πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα. Ε, ε, τον Σεπτέμβριο επίσης είχαμε μια πολύ συγκεκριμένη ε, περίπτωση διαφάνειας, μια επιστολή από την ΕΚΤ στον Υπουργό Οικονομικών της Ιρλανδίας τον Οκτώβριο. Έγινε παράλληλη λοιπόν έρευνα. Κάποια από τα κράτη-μέλη είχαν και αυτό το δικό τους διαμεσολαβητή που συμμετείχε. Εδώ είναι τα νούμερα για πέρυσι, δεν έχουν αλλάξει και πολύ. Βοηθήσαμε περίπου 23.000 ε, πολίτες, ε, κυρίως ε, μέσω του interactive οδηγού στο διαδίκτυο. Και οι καταγγελίες που είχαν κυρίως είχαν να κάνουν με τη δική τους εθνική διοίκηση. Τους βοηθήσαμε λοιπόν να στείλουν την καταγγελία τους στην κατάλληλη αρχή, είτε το δικό τους ε, διαμεσολαβητή, είτε την Επιτροπή Αναφορών ή ε, σε κάποιον από τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται με αυτές τις έρευνες. Όλοι όμως βοηθούνται, όλοι παίρνουν μια ατομική απάντηση. Όσον αφορά τώρα τις επίσημες έρευνες που ξεκίνησαν. Ξεκινήσαν 425 τέτοιες ακροματικές διαδικασίες το 2014 και, οι 400 έχουν, και 400 έχουν κλείσει. Για άλλη μια φορά λοιπόν τα τελευταία χρόνια δεν αλλάζουν και πολύ τα νούμερα. Εδώ βλέπετε τις βασικούς ε, θεσμούς με τους οποίους ασχοληθήκαμε. Δηλαδή όσον αφορά στις καταγγελίες, ε, προφανώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ε, αυτή που έχει το κομμάτι του λέοντος, γιατί ε, όχι επειδή είναι ιδιαίτερα κακή, αλλά επειδή ε, όπως καταλαβαίνετε έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στη ζούγκλα και γι' αυτό οι περισσότεροι πολίτες την αυτήν τους καταγγελίες τους 47 οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρυθμιστικές αρχές, άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν δουλειά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θεωρούν ότι ήταν άδικη διαδικασία επιλογή του έρχονται σε εμά, ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. οι καταγγελίε εκεί έχουν να κάνουν με διοικητικά ζητήματα και με τι αποστολέ που έγιναν σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρόμοιες περιπτώσεις και φυσικά η Όλαφ. Ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Πάταξη της Απάτης. Τώρα για τη συμμόρφωση του 2013 αυτή είναι η πίτα που βλέπετε. Έχουμε τις, ε, την έκθεση, ε, που, τον απολογισμό που θα γίνει για την συμμόρφωση σύντομα. 80% συμμόρφωση, 20% μη συμμόρφωση. Για άλλη μια φορά, όπως έχω πει πολλές φορές, ε, επαναλαμβάνω και τώρα ότι θέλω να αυξηθεί αυτό το νούμερο. Διότι ε, στις περισσότερες περιπτώσεις στους διαμεσολαβητές είναι 90% η συμμόρφωση. Δεν είναι και τόσο δύσκολο, πιστεύω, να πάμε στο 90% λοιπόν να συνεργαστούμε με τα θεσμικά όργανα. Τώρα, το βασικό ζήτημα, έλλειψη διαφάνειας. Ε, ο κόσμος προσπαθεί να βρει αρχεία και δεν έχει πρόσβαση ή τους ε, αρνούνται την πρόσβαση, οπότε προσφεύγουν σε εμά. Διαφάνεια όσον αφορά στις ομάδες πίεσης να δώσουμε κάποια πίστοση στην Κομισιόν για τις ε, προσπάθειες που έχει κάνει σε αυτόν εδώ τον τομέα. Υπάρχει η πρωτοβουλία για την διαφάνεια που ξεκίνησε από την Κομισιόν φέτος και έχουμε όλο και περισσότερες πληροφορίες για τις συνεδριάσεις που κάνουν οι επίτροποι και τα επιτελεία τους και οι γενικοί διευθυντές με ε, ανθρώπους που έρχονται για να ασκήσουν πίεση σε αυτούς ή να τους μιλήσουν απλώς. Ε, εξαρτάται επίσης από τον ίδιο το λομπίστα θα θέλει να δημοσιευτεί το όνομά του. Πολλές φορές έχουμε το όνομα της οργάνωσης, αλλά δεν έχουμε τον εκπρόσωπο ως όνομα, τον οποίο δηλαδή συνάντησε ο Επίτροπος. Πολλέ φορέ ε, η Κομισιόν λέει ότι αυτό είναι ένα αίμα προστασία προσωπικών δεδομένων. Εγώ δεν το δέχομαι τόσο, διότι θα μπορούσε απλώ η Κομισιόν να ε, λέει ότι από τη στιγμή που κάποιος ζητά συνάντηση με την Κομισιόν θα πρέπει να δημοσιεύεται και το όνομά του, να το δέχεται αυτό. Επίσης, το ίδιο πρέπει να γίνεται και για αυτούς που είναι και σε χαμηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας, γιατί το lobbying δεν γίνεται μόνο με τους επιτρόπους, γίνεται και στα χαμηλότερα επίπεδα και δεν είναι πρόβλημα το λόμπινγκ, απλώς καλό θα είναι ε, ποιος έχει, να ξέρουμε ποιος έχει συναντηθεί με ποιον όταν προωθείται ας πούμε ένα ε, νομοθετικό ε, έγγραφο, καλό είναι να γνωρίζουμε πώς προέκυψε. Περιμένουμε την απάντηση της Επιτροπής, ειδικά όσον αφορά μια συγκεκριμένη σύσταση που έκανα και σας την έχω ξαναπεί νομίζω, συγκεκριμένα όταν ανώτατοι αξιωματούχοι φεύγουν και πάνε στον ιδιωτικό τομέα, Πολλές φορές μπορεί να υπάρχει σύγκρουση σε σχέση με τη δουλειά που έκαναν προηγουμένως στην Κομισιόν. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει δημόσια πρόσβαση σε ένα μητρό όπου θα βλέπουμε τα ονόματα, τον τρόπο εργασίας, τι έκαναν με την Επιτροπή έτσι ώστε να γνωρίζουμε τυχόν περιορισμούς που υφίστανται για την εργασία τους στον ιδιωτικό τομέα και η Κομισιόν και όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να δεσμεύονται να δίνουν πληροφορίες γι' αυτό. Αυτό που είπε η Κομισιόν ήταν ότι στα τέλη του έτου ε, θα μα δίνουν κάποιες ε, αναφορές για αυτό το θέμα, να δούμε ποια θα είναι η μορφή των αναφορών. Επίσης, οι δεδομένων. Έχουν γίνει πολλές ε, μορφές συναντήσεων μεταξύ Ευρωπαϊκών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ατόμων, εταιριών κτλ. Έτσι λειτουργεί το πράγμα. Αυτό που εγώ λέω είναι ότι η πρόσβαση μάλλον δεν είναι τόσο ισορροπημένη. Πρόσφατα έγραψα στον πρόεδρο του ΕΚΤ, τον Μπάριο Ντράγκη, για να του μιλήσω για μια ιδιωτική συνάντηση που είχε γίνει στο Λονδίνο. Ένας εκτελεστικός διευθυντής της ΕΚΤ είχε ε, δώσει ευαίσθητες πληροφορίες ε, σχετικά με την αγορά και ήθελα να μου εξηγήσει ο πρόεδρος της ΕΚΤ τι ακριβώς είχε συμβεί. Ήταν διοικητικό το θέμα. Ε, η απάντηση του κύριου Ντράγκη ήταν ότι αυτός ε, και το Συμβούλιο θα ε, δουν τώρα ε, ποια είναι τα πρωτόκολλα συνάντησης με ανθρώπους από τον ιδιωτικό τομέα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και σε αυτό το τομέα. Τώρα, στρατηγικές έρευνες. Το, σας, σας το είπα και πριν, έχουμε δώσει περισσότερη έμφαση σε αυτό. Είμαστε ένα μικρό γραφείο, 65 άτομα και είναι ηθική μου υποχρέωση να κάνω τη μέγιστη χρήση των ε, διαθέσιμων πόρων. Και εγώ προσωπικά ασχολούμαι με τις καταγγελίες ε, και το γραφείο μου ε, πραγματικά θα είναι πιο χρήσιμο θεωρώ αν αντιμετωπίσει τα συστημικά προβλήματα γιατί έτσι αυτό θα μπορέσει να λύσει τα προβλήματα και, πολλά, και πολλών ατόμων ξεχωριστά. Ένα, μία από τις μεγάλες πρωτοβουλίες που ξεκίνησε πέρυσι ήταν ε, αυτή για τη διαφάνεια με, στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Όλοι το γνωρίζετε αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλοι παράγοντες ε, της κοινωνίας των πολιτών ήταν ιδιαίτερα ενεργοί σε αυτό το τομέα. Ως αποτέλεσμα της δικής σας δουλειάς και της δικής μου δουλειάς, η Κομισιόν τώρα είναι όλο και περισσότερο πιο προμηθής όσον αφορά στις εκθέσεις ε, που βγάζει το διαδίκτυο, εκ των προτέρων δηλαδή προσπαθεί να λύσει προβλήματα. Φτάνουμε λοιπόν στο επίπεδο να έχουμε τελικά ένα ολοκληρωμένο κείμενο ε, για μια σχέση, για μια συμφωνία που ενδεχομένως έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλέ φορές υπάρχει χάσμα μεταξύ αυτού που θέλει να ε, δημοσιεύσει η πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό που τελικά ε, πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές ε, δεν συνάδουν αυτά με την, τον κανονισμό 1049 και πολλές φορές ε, υπάρχουν αντιρρήσεις οι οποίες ε, από την πλευρά των ΗΠΑ πολλές φορές οι οποίες πρέπει να αξιολογηθούν. Τώρα, η Frontex. Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν για κάποιες από τις έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με την Frontex. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια κοινή ακρόαση με αυτή την Επιτροπή και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ Όσον αφορά μια συγκεκριμένη έκθεση που προήλθε από τον προκάτοχό μου, την οποία ψηφίσαμε στο Κοινοβούλιο και πρόκειται για μια συγκεκριμένη σύσταση. Η σύσταση, η Frontex, να έχει έναν μηχανισμό καταγγελιών όπως και τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε όσοι θεωρούνται ότι αδικήθηκαν ή έχουν παράπονα, να μπορούν να έχουν κάπου να προσφύγουν. Ας πούμε, ε, κατάχρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή παραβίαση δικαιωμάτων ελεύθερης έκφρασης. Αυτό μπορεί να συμβεί σε πολλά κρατημέλη. Από τη στιγμή που υπάρχουν όμως Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί θα μπορούσαν να είναι το κεντρικό σημείο μέσα από το οποίο θα μπορούσαν να φιλτράρονται οι καταγγελίες του κόσμου. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει μια έκθεση γι' αυτό. Επίσης ε, για τις αναγκαστικές επιστροφές ε, των ε, μεταναστών είναι ένα τεράστιο θέμα. Άνθρωποι που διασχίζουν τη Μεσόγειο και έρχονται στην Ευρώπη. Πολλοί άνθρωποι έχουν πνιγεί στην προσπάθεια αυτή. Έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο πολύπλοκο είναι αυτό το ζήτημα. Έτσι λοιπόν πέρυσι κάναμε μια έρευνα σχετικά με τις ε, ε, επιχειρήσεις επιστροφής που συντονίζει η Frontex σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, αν η Ισπανία έχει αποφασίσει ότι κάποιοι αιτούντες άσυλο πρέπει να φύγουν από την χώρα, η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Frontex ε, συντονίζει τις πτήσεις, κοινέ πτήσεις, οι οποίες φέρνουν τον κόσμο ξανά στην χώρα προέλευσής του. Στην... Στον τομέα λοιπόν αυτό, η Frontex μας έδειξε ένα βίντεο με τις πτήσεις αυτές ε, που πραγματικά γέννησε πολλά ερωτήματα στο μυαλό μου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία τους σε αυτές τις πτήσεις. Ζήτησα λοιπόν από τους ε, ε, διαμεσολαβητές στα κράτη-μέλη να κάνουμε μια παράλληλη έρευνα για αυτό το ζήτημα και πραγματικά με ενθουσιασμό δέχτηκαν την πρόσκλησή μου. Πολλοί λοιπόν διαμεσολαβητές από την Ισπανία, την Ολλανδία, την, Πολωνία, όλοι κάνουν και τη δική τους έρευνα για αυτό το θέμα και σύντομα θα γίνει μια συνάντηση έτσι ώστε ε, να δούμε τι γίνεται και επίσης να εκδοθούν και οι εθνικές εκθέσεις. Το μήνυμα, η σύσταση που έδωσα στις Frontex είναι ότι πρέπει να εναρμονιστούν οι τρόποι με, τον οποίο, με τους οποίους αντιμετωπίζονται π.χ. οι έγκυες γυναίκες ή τα παιδιά που επιστρέφουν στις χώρες τους. Πρέπει να υπάρχει μια σειρά συμφωνημένων κανόνων και να μην εξαρτώμαστε κάθε φορά από τα στάνταρ της κάθε χώρας. Η Frontex δηλαδή να μην έχει ένα ε, εναρμονισμένο πλαίσιο προτύπων υψηλού επίπεδου. Άλλη μια έρευνα που έκανα ήταν για αυτό το θέμα που βλέπετε στην οθόνη σας, ε, δηλαδή την ε, πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, το θέμα δεν ήταν αν θα έπρεπε να δέχεται η Κομισιόν αυτές τις πρωτοβουλίες, αλλά θα πρέπει να σκέφτεται πώς ακριβώς θα προσεγγίζει τους ανθρώπους που μπήκαν στον κόπο να ξεκινήσουν μια τέτοια πρωτοβουλία. Πώς λοιπόν θα τους απορρίψει ενδεχομένως την πρωτοβουλία τους, πώς να εξετάζει την ε, πρωτοβουλία που έχει συλλέξει ένα εκατομμύριο υπογραφές και ούτω καθεξής. Ο κύριος Τίμερμαν, ο πρώτος ε, αντιπρόεδρος, κατανοεί από την Κομισιόν, εκ μέρους της Κομισιόν, ότι σε κάποιες περιπτώσεις η απάντηση της Κομισιόν ήταν πολύ νομικήστικη. Έπρεπε να υπάρχει μια πιο πολιτική απάντηση. Εγώ λοιπόν ενδιαφερόμουν κυρίως ε, για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σωστά οι πρωτοβουλίες αυτές, πώς να επικοινωνούν δηλαδή με τον κόσμο με τέτοιο τρόπο ώστε να ε, να αποφεύγεται η λάθος μεταχείρισή τους. Τώρα αυτό το θέμα δεν σχετίζεται άμεσα με το 2014. Είναι μια έρευνα ιδέας πρωτοβουλίας που θα ξεκινήσει σύντομα σχετικά με την διαφάνεια των διαδικασιών του τριμερούς διαλόγου. Τους τελευταίους 18 μήνες δεν είχαμε κάποιες επίσημες ε, καταγγελίες, αλλά είχαμε ένα διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, τους ε, προβουλευτές ε, και πολλοί ανησυχούν για την έλλειψη διαφάνειας σε αυτή τη διαδικασία. Πολλοί λένε ότι τους αποκλείουν από την νομοθετική διαδικασία που θα έπρεπε να είναι πολύ πιο διαφανής. Οπότε δεν πρέπει να κοιτάμε ε, ποια είναι τα σωστά ή τα λάθος. Υπάρχουν ε, πολλές ε, αποφάσεις οι οποίες σωστά βγαίνουν από τον τριμερή διάλογο. Εμείς απλώς θέλουμε να χαρτογραφήσουμε τη διαφάνεια στον τριμερείς διαλόγους και ζήτησα από το Συμβούλιο, την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο να μας δώσουν κάποιες γενικές πληροφορίες καταρχάς για να δούμε τι είναι αυτό που είναι πιο ορατό, τι δεν είναι διαφανές και ποια είναι τα διάφορα στάδια της διαδικασίας. Δεν κοιτάμε λοιπόν τις πολιτικές, τα πολιτικά παζαρία, κοιτάμε λίγο πολύ τι γίνεται σε επίπεδο διαφάνειας. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που μας παρουσιάσατε αυτήν την τόσο ενδιαφέρουσα έκθεση την οποία συστήνω σε όλους μας. Να τη διαβάσετε. Και τώρα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους για ερωτήσεις. Ο κύριος Βαλέσα πρώτος. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ράιλ. Κάθε φορά είναι μεγάλη χαρά μας όταν σας ακούμε γιατί μας εμπνέεται και ιδίως αυτά που λέτε μας δίνουν και μας ε, ελπίδα και κουράγιο για να βελτιώσουμε και τη συμμετοχή των πολιτών ε, Έχω όμω ε, κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για μια ακόμη φορά περισσότερα ήταν ε, τα αιτήματα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά χωρίς να διακινδυνεύσουμε την ε, δημόσια ασφάλεια και τη διαπραγματευτική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, τι είδου προκλήσεις εσεί έως το 2014. Σε ό,τι αφορά τη μη συμμόρφωση των θεσμικών οργάνων τη Ένωση στι προτάσει σα. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Με βάση τα στοιχεία τη ετήσια έκθεση, βλέπουμε σταθερή ε, μείωση των καταγγελιών εκτός ε, της εντολής ε, εκτός πλαισίων εντολής ε, της διαμεσολαβητρίας. Γιατί έχουμε αυτή τη σημαντική θετική μείωση. Τρίτη ερώτηση για την ίδια την έκθεση στην ιστοσελίδα μόνο στα αγγλικά διατίθεται. Πάντα θέτω το σχετικό ερώτημα. Προβλέπετε μετάφραση της ετήσιας έκθεσης σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Παραλαμβάνω δηλαδή και το περσινό μας αίτημα. Τέλος. Έχουμε πολλές καταγεγραμμένες ε, καταγγελίες ε, που μεταφέρονται σε άλλα μέλη του δικτύου του Ευρωπαίου Μεσολαβητή. Υπάρχουν μηχανισμοί για την παρακολούθηση, για τη συνέχεια που δίνεται σε αυτή τη μεταφορά, των, ε, τη διαβίωση των καταγγελίων, ώστε να εξεταστούν πράγματι. Ο κύριος Τέρι Κάμπρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Ρέλη που είστε εδώ σήμερα και που μας παρουσιάσετε το έργο σας. Σύντομο το ερώτημά μου και πολύ συγκεκριμένο. Λέτε ότι έχουμε 80% συμμόρφωση. Τι γίνεται με το 20% της μη συμμόρφωσης. Τι γίνεται. Τίποτε. Τίποτε δεν γίνεται. Με αντιδρούν στις δικές σας υποδείξεις. Δεν κάνουν τίποτε. Δεν απαντούν, δεν ανταποκρίνονται. Δεν γίνεται τίποτε. Γιατί αυτό είναι σημαντικό. Για τη δική σας ε, την εξουσία, μπορώ να το πω έτσι, και το κύρος σας ως αρχής. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο στον καταλογό μου. ο κύριο Γιάννη. Äh, Μια σύντομη ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ε, ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστούμε και για την υποστήριξη σχετικά με το θέμα της διαφάνειας ε, στα πλαίσια του TTIP. Να πω ότι έχουμε καταφέρει από κοινού βελτιώσεις και στο θέμα των ε, ευρωβουλευτών ε, που πραγματικά συνεισέφεραν. Ε, ήμασταν και οι ίδιοι τόσο μη ικανοποιημένοι εξ αρχής, διότι δεν είχαμε πρόσβαση στα έγγραφα. Τώρα έχει βελτιωθεί αυτό, περάσαμε αυτό το σκοτεινό δωμάτιο σε ένα δωμάτιο που μπορούμε να δούμε πια. Και μετά έχουμε ε, καταφέρει πλέον να συζητούμε με τους πολίτες το θέμα της TTIP. Τώρα, για το θέμα της διαφάνειας, ε, πάντοτε υπάρχει αυτό το θέμα των προσωπικών δεδομένων. Ε, χτυπάμε πάνω σε αυτό το θέμα. Και η διαφάνεια πρέπει να έχει δηλαδή κάποια συγκεκριμένα όρια, ε, λέγεται. Και ε, υπάρχει και αυτή η ζυγαριά. Ε, που πάντοτε ζυγίζουμε ποιο είναι καλό και ποιο είναι κακό, τι είναι το λιγότερο καλό και το λιγότερο κακό. Ε, πολλές φορές τα προσωπικά δεδομένα είναι στην αντίθετη πλευρά της διαφάνειας. Όπως και να έχει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το θέμα της διαφάνειας στην DZIP. ακόμα και τα μη, ε, περί, τα μη αμφιλεγόμενα ζητήματα γίνονται αμφιλεγόμενα όταν δεν υπάρχει διαφάνεια και γι' αυτό ευχαριστούμε για τη διαφάνεια. Έχουμε έτσι τη δυνατότητα να έχουμε δημοκρατικά νομιμοποιημένες αποφάσεις. Ευχαριστώ. Μίσης Βαλίνα. κυρία Βαλίνα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα Ουσιαστικά δεν έχω κάποια ερώτηση, κυρίως ε, θέλω να συγχαρώ για την πολύ χαραλή αυτή έκθεση στην ε, κυρία βίτρια Αυτό μας ζητά ε, κοινή γνώμη, μα ζητά διαφάνεια, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και πράγματι ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνειας, ε, οι επισκέψεις αυτές των ομάδων πίεσης που πολλές φορές κανείς υποκύπτει πιο εύκολες πιέσεις των ομάδων αυτών και όχι στους ε, πολίτες. Άλλωστε όμως πρέπει, να, πρέπει όμως να ξέρουμε, θα σου πω, δεν τους έχει εκλέξει κανείς ε, τους λομπίστες εννοώ. Λοιπόν, πολλά από τα θέματα που θίξατε, τη μεταπίδηση από το δημόσιο στον τομέα, αυτά revolving doors πράγματι ε, και στη χώρα μου την Ισπανία ε, έχουμε ε, τέτοια παραδείγματα ε, και πρέπει να βάλουμε τροχοπέδι στο φαινόμενο αυτό διότι στερεί από τους θεσμούς και από την πολιτική και τους πολιτικούς την αξιοπιστία τους. Και τελικά τι είδαμε και στις τελευταίες ευρωεκλογές να έχουν ψηφίσει λιγότερο από το 50% των πολιτών. Μια ερώτηση όμως να σας ε, υποβάλω. Σε ποιο βαθμό δίνει σημασία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις του θεσμού του Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή. Ευχαριστώ κυρία Πιτέρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η έκθεσή σας ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Έχω μία ερώτηση. Εγώ άρχισα να ενδιαφέρομαι ιδιαίτερως για ένα στοιχείο αυτής της έκθεσης κυρίως ότι δεν υπάρχει συμφωνία για παροχή πληροφοριών και για γνωστοποίηση των ονομάτων όσων έρχονται σε επαφή με επαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν την καταλαβαίνω αυτή την επιχειρηματολογία και είναι κάτι που αντιμετωπίζω ε, από καιρό εις καιρών. Δεν είναι όμως κατηδίαν συναντήσεις αυτές. Είναι επίσημες, δημόσιες και ε, επηρεάζουν το σχεδιασμό πολιτικής ως προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών με τρίτες χώρες. Οι υπάλληλοι αυτοί, οι άνθρωποι αυτοί απλώς ε, κάνουν τη δουλειά τους. Δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από την προστασία των δεδομένων και η επιχειρηματολογία αυτή είναι εκτός ε, θέματος, διότι η διαφάνεια θα πει ότι πρέπει να έχουμε γνώση για όλα τα μέρη που συμμετέχουν σε μια διοικητική διαδικασία, διότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε έλλειψη ισορροπίας. Οπότε ή θα είμαστε πλήρως διαφανείς είτε καθόλου. Θέλω λοιπόν να μου πείτε ποια είναι η λογική. Η λογική πέραν αυτής της επίσημης ε, δικαιολογίας που χρησιμοποιείται. Ποια είναι η λογική του να αποκρύπτονται αυτές οι πληροφορίες. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι ανεξάρτητα άτομα. Είναι άνθρωποι υπάλληλοι που εκπροσωπούν έναν επίσημο φορέα. Και επιπλέον πολλές φορές έχουν να κάνουν με δημόσιες υποθέσεις, με, κοινά, με τα κοινά όταν ε, συζητούν αυτές τις αντίστοιχες. Ευχαριστούμε κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε για την ε, δουλειά σας, Έμιλη είναι εντυπωσιακή και θα δούμε πώς θα επιβιώσετε από όλη αυτή τη φοιτεία στην Δανία. θυμάμαι να παρουσιάζεται ο διαμεσολαβητής σαν ένας Δαβίδ που είχε να τα βάλει με έναν Γολιάθ. Είσαστε λοιπόν όντω μια μικρή υπηρεσία που έχετε να τα βάλετε με μεγάλε δυνάμει. Ε, τώρα, η έκκλησή σα για διαφάνεια και για του τρεμερεί διαλόγους όλος ιδιαίτερο. Ξέρετε ότι εγώ είμαι ο Ναφανδόν υπέρ της ε, διαφάνειας και εδώ υπάρχει πραγματικά έλλειψη ισορροπία, διότι το Συμβούλιο δεν την θέλει. Όταν λέτε λοιπόν πως είστε εκτεθειμένοι στους, ε, στις ομάδες πίεσης και εδώ νομίζω ένα πράγμα πρέπει να είναι σαφές ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μπορεί να αποδυναμωθεί δραματικά το κοινοβούλιο εάν έχουμε πληθέσεις από όλες τις πλευρές από ομάδες πίεσης και λόμπι Και εδώ ίσως τελικά να έχουμε ένα μεγαλύτερο παράγοντα ασφάλειας στους τριμμένους διαλόγους αν τα πάντα δεν είναι δημοσιοποιημένα. Και το Συμβούλιο δεν θέλει κάτι τέτοιο. Οπότε θα θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό. Διότι κάπως έτσι σχολιάζεται το θέμα στην ομάδα μου. Thank you very much. Ευχαριστούμε και έτσι ολοκληρώνει το κατάλογο των ομιλητών. Όχι τώρα και η κυρία Μπεσέρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Ρέλη, σας ευχαριστούμε που έρχεστε για μια ακόμη φορά. Πραγματική χαρά να σας ακούμε. Έχει, έχετε αναλάβει τα καθήκοντά σας ε, για πέντε χρόνια. Έρχεται έρθει δύο φορές στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να μας πείτε κάποια πράγματα σε σχέση με τις θεσμικές σχέσεις ε, με τα όργανα. Έχει αλλάξει καθόλου τη δουλειά σας το γεγονός ότι η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει αυτή τη ε, στιγμή έναν ε, αντιπρόεδρο με πολλές αρμοδιότητες, τον κύριο Τίμερμανς και στο χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνονται οι πολίτες στα θέματα της αργένειας. Σας το ρωτώ αυτό διότι η στενή συνεργασία αυτό το, στενό, το πλαίσιο στενής, στενής συνεργασίας ε, που δημιουργήθηκε μεταξύ του Γραφείου του Διαμεσολαβητή και της Επιτροπής μας ουσιαστικά ε, συνεπάγεται το να δώσουμε υπηρεσία στον πολίτη. Είμαστε ίσως οι δύο όψεις του διονομίσματος και υπάρχει και μια τρίτη όψη, οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλάζει τίποτα στο δικό σας έργο ύπαρξη αυτού του νέου αντιπροέδρου. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας ευχαριστήσω και εγώ κυρία Ράιλι και να σας συγχαρώ για αυτή την έκθεση που είναι πραγματικά μία ε, έκθεση που μας εμπνέει και μας ενθουσιάζει. Η προσέγγιση που βγαίνει, ε, το μήνυμα που βγαίνει είναι ότι είστε πραγματικά στο πλευρό των πολιτών, ότι διευκολύνεται την επίλυση των προβλημάτων τους. Είμαστε υπερήφανοι λοιπόν που μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί σας και να βρούμε βιώσιμες λύσεις σε αυτά τα συστηματικά προβλήματα, ζητήματα όπως η διαφάνεια, πράγματα που θέλουμε πραγματικά να συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες μαζί σας. Τώρα, αυτό που είπαμε για το ότι θέλετε να μην είμαστε τόσο νομικίστικοι στην ε, προσέγγιση μας όσον αφορά ας πούμε τις πρωτοβουλίες των πολιτών πραγματικά ε, είμαστε ανοιχτοί ακόμα και στις πρωτοβουλίες που απορρίπτονται γιατί η πολιτική ουσία και η προσπάθεια που έχει επενδύσει ο κόσμος σε αυτές τις πρωτοβουλίες το να βρει κανείς σχεδόν ένα εκατομμύριο υπογραφές καταλαβαίνετε είναι κάτι που πρέπει να το εκμεταλλευτούμε να μπούμε σε μια συζήτηση, σε διάλογο μαζί με αυτούς τους ανθρώπους Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ που μπορέσατε να μοιραστείτε μαζί μας κάποιες στιγμές και τώρα σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που σας ετέθησαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για τα ευγενικά σας λόγια. Το εκτιμώ και εγώ και οι συναδελφοί μου. Ευχαριστώ κύριε Βαλέσα για τις ερωτήσεις σας. Να πω πρώτα στο κομμάτι της μετάφρασης, τη στιγμή που μιλάμε, τα πάντα μεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έχουμε συμβάσεις για όλα αυτά. Αύξηση της διαφάνειας. Το είπα και πριν. Νομίζω ότι υπάρχουν εξαιρετικές ευκαιρίες ε, τα επόμενα τέσσερα χρόνια να κάνουμε τη διαφάνεια πιο μεγάλη σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι υπάρχει μεγαλύτερη απέτηση από την πλευρά των πολιτών ε, που ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια, ειδικότερα μετά την ύφεση και την οικονομική κρίση που έχει επηρεάσει τόσο κόσμο. Δεν είναι απλώς θυμωμένοι. Απαιτούν να δουν πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, πώς λειτουργούν οι θεσμοί. Ζητούν απαντήσεις και η Κομισιόν το ζητά αυτό, μιλά πολύ για τη διαφάνεια, το έχει ενσωματώσει, έχει βγάλει την ε, διαφάνεια στο προσκήνιο, στη μεγαλύτερη αξία που ε, πρεσβεύει και πρέπει ε, να συνταχθούμε με αυτό. Τώρα για πιο τεχνικά ζητήματα, επειδή από τη στιγμή που έγινα ομπουτσμαν και πριν από αυτό, υπήρχε μεγάλη συζήτηση για την αναθεώρηση του κανονισμού 1049. Δεν ξέρω που ακριβώς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, αλλά προφανώς αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά στο Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα. Αυτά θα το εξετάσουν. Τώρα, για τις ε, καταγγελίες σχετικά με τις θητείες, ε, να πω ότι οι συνάδελφοι στο Μητρό, στο γραφείο μου, έχουν ε, εργαστεί πολύ σκληρά τα τελευταία χρόνια για να μπορέσουν να μειώσουν τον αριθμό των ανθρώπων που, λαμβάνουν μια που δεν λαμβάνουν απάντηση. Έχουμε αυτό τον interactive οδηγό ο οποίος ε, βοηθά να δει κανείς αν πρέπει να απευθυνθεί στον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή ή, ε, διαμεσολαβητή ή όχι. Ο προκάτοχός μου, ε, ο κύριος Διαμαντούρος, το είχε θέσει αυτό το πρόβλημα, το ήξερα λοιπόν πριν γίνω διαμεσολαβήτρια και από ό,τι φαίνεται η προσπάθεια που κάναμε αποδίδει. Τώρα για τη μεταφορά των καταγγελιών, ποιος το ρώτησε αυτό, μισό λεπτό. Ναι, Όντως, γίνεται ένα follow-up, όχι με επίσημο τρόπο, αλλά όταν γίνεται κάποια μεταφορά, υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ εμού και του ομολόγου μου στο κράτος μέλος που έχει αναλάβει την καταγγελία. Είτε συναντιόμαστε σε κάποια σεμινάρια, είτε μιλάμε μέσω διαδικτύου. Γενικά όμως υπάρχει επικοινωνία παρακολουθούμε το θέμα. Δεν είναι εδώ ο συνάδελφος. Εντάξει, δεν πειράζει. Το 20% των, ε, της μη συμμόρφωσης των καταγγελιών που δεν γίνονται αποδεκτές. Κοιτάξτε, και εγώ το εξετάζω αυτό. Εξ αρχής είπα και το είπα και στις ακροάσεις μου για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ότι θέλω να ερευνήσω τι γίνεται και να μειώσω αυτό το ποσοστό. Προσπαθώ να γίνω λίγο πιο ευθύνη με, το, με τα θεσμικά όργανα. Κάνω περισσότερες ε, συστάσεις, δεν δίνω κατευθυντήριες γραμμές απλώς. Ε, είμαι λίγο πιο επίμονη. Συνεργάζομαι όμως μαζί τους και πιο έντονα, πιο εντατικά και είχα συναντήσεις με ανώτατους αξιωματούχους στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν που ασχολούνται με την διαφάνεια και έχουμε με πολύ συνεργατικό τρόπο συζητήσει τα συγκεκριμένα θέματα στα οποία διαφωνούμε. Αυτό κάνουμε. Στην ουσία μιλάμε και έχουμε επαφές. Όχι μόνο στο υψηλό επίπεδο, αλλά και στο χαμηλότερο επίπεδο στους ανθρώπους που συνεργάζονται με τους δικούς μου, ε, με το δικό μου γραφείο, του συναδέλφους μου κύριε Γιάννη, για την προστασία των δεδομένων. Το λέω συχνά ότι με εξέπληξε όταν ήρθα στην Ευρώπη εντό εισαγωγικών το γεγονός ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων πολύ συχνά χρησιμοποιείται ως ε, δικαιολογία, ως πρόφαση για να μην υπάρχει διαφάνεια. Αυτό δεν θέλω να υφίσταται. Οι κανονισμοί πάντοτε μπορούν να έχουν ε, το δημόσιο συμφέρον πάντα στο πρώτο πλάνο, ακόμα και όταν διακυβεύονται τα προσωπικά συμφέροντα. Ακόμα και σε κάποιες από τις υποθέσεις που σας έχω παρουσιάσει, μία ας πούμε που έχει να κάνει με τη μεταπίδηση από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, η πρόταση που έκανα στην Κομισιόν να βάλουν ένα μητρό δημοσίως ε, προσβάσιμο στο ίντερνετ ε, που να μπορεί κανείς να βλέπει τι ακριβώς γίνεται. Ακόμα και σε αυτό το θέμα μας επανέλαβαν το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων. Βέβαια, να συγχαρούμε την Κομισιόν για την διαφάνεια σε επίπεδο συναντήσεων ε, ε, επιτρόπων και επιτελείου των επιτρόπων και γενικών διευθυντών. Τώρα βέβαια ζητούν από τους ανθρώπους να δώσουν την συγκατάθεσή τους για το να δημοσιευτεί το όνομά τους. Όμως δεν θεωρώ ότι αυτό είναι σωστό. Αυτό πρέπει να είναι μέρος ε, του δημοσίου δικαίου και των κανονισμών. Τώρα για το revolving doors, την μεταπίδευση από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, νομίζω ότι Αυτά τα ζητήματα τα βλέπουμε πολλές φορές στον τύπο και κατανοούμε πόσο καταστρέφουν την εικόνα των θεσμών, την εμπιστοσύνη του κόσμου. Και βλάπτουν φυσικά και τους πολύ καλούς υπαλλήλους ε, στο, στα θεσμικά όργανα. Έχω συζητήσει λοιπόν με πολλούς από τους ανθρώπους που τελικά υποστηρίζουν αυτές τις προτάσεις που έχω κάνει για τέτοια ζητήματα, διότι οι περισσότεροι είναι περήφανοι για τη δουλειά που κάνουν και βλέπουν ότι η δουλειά τους βλάπτε όταν υπάρχουν κάποιοι που δεν συμπεριφέρονται σωστά και δεν έχει γίνει και σωστή, ε, σωστός έλεγχος ε, της συμπεριφοράς αυτής. Κυρία Πιτέρα, ναι, όντως έχουμε συζητήσει το θέμα των συναντήσεων με την Κομισιόν. Συμφωνώ ότι είναι σημαντικό κομμάτι της διαφάνειας να ρωτά κανείς ε, ποια είναι η λογική ε, που ε, επιζητά να αποκρύπτονται κάποιες συναντήσεις. Ίσως είναι πολιτισμικό το ζήτημα. Στα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα ίσως να μην έχει κανείς μεγάλη δυσκολία να αποδέχεται να μαθαίνει τι γίνεται με το δημόσιο χρήμα. Σε άλλες κουλτούρες αυτό δεν είναι τόσο αποδεκτό. Γενικά όμως θεωρώ ότι η κουλτούρα, ο πολιτισμός πηγαίνει προς μια συγκεκριμένη κατάθεση, κατεύθυνση. Κατά τη γνώμη μου είναι μια μορφή εξέλιξης και νομίζω ότι πάντοτε μέσα στα πλαίσια μιας θητείας βλέπουμε σταδιακές βελτιώσεις σε αυτά τα θέματα. Τώρα, για το σχόλιο σχετικά με το μικρό γραφείο έναντι του μεγάλου γραφείου να πω ότι ναι, το δικό μου γραφείο είναι μικρό, αλλά έχουμε και το κοινοβούλιο που είναι ένα μεγάλο γραφείο και σας έχω μαζί μου. Ε, το να έχεις 65 άτομα στο γραφείο σου είναι κάτι που το καθιστά μικρό. Όμως μπορεί να έχει κάποια ε, εξουσία, κάποιο βάρος και πολλές φορές έχω πει πόσο σημαντική είναι η σχέση μεταξύ μας ε, δηλαδή του γραφείου μου και του Κοινοβουλίου. Πολλές φορές έχω επαναλάβει πόσο σημαντική είναι η συνεργασία μας και πολλές φορές καλωσορίζω τις πρωτοβουλίες κυρίας Βίκστρομ για αυτό το θέμα. Τώρα, για τη χαρτογράφηση που θα γίνει για τους τριμερείς διαλόγους, να πω ότι αν υπάρχει και υπερβολική διαφάνεια και οι λομπίστες βλέπουν τι σκέφτεται ο καθένας, τελικά θα τρομοκρατηθούν από τους ανθρώπους που τελικά θα σειρεύσουν για να περάσουν την άποψή τους. Βέβαια, ε, η διαφάνεια δεν είναι και για να βλάψει, ούτε και για δικούς της σκοπούς. Απλώς για να έχουμε διαφάνεια δηλαδή. Αυτό που λέω συνήθως είναι ότι πρέπει να δούμε τι υπάρχει, τι γίνεται και ό,τι μπορεί να δημοσιευτεί, να δημοσιευτεί. Ε, ένα καθεστώς διαφάνειας είναι λανθασμένο ή δεν εφαρμόζεται σωστά αν τελικά με την ε, πρόορη πολλές φορές ε, ή μη αποκάλυψη των αρχείων βλάπτεται ο κόσμος, το δημόσιο συμφέρον. Συγκεκριμένα θα εξετάσουμε κάποιους συγκεκριμένους ε, τριμερείς διαλόγους, όχι όλους, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Έχουμε επιλέξει δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις για να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να δώσουμε σε επίπεδο διαφάνειας. Τώρα το ερώτημα σχετικά με το αν άλλαξε η δουλειά μου σχετικά με τον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς και τη διεύρυνση του ρόλου του για τα δικαιώματα των πολιτών, να πω ότι βοήθησε. Γιατί έχουμε αναγκαστεί να συζητάμε περισσότερο. Είμαστε στην ίδια πλατφόρμα. Και αυτός και εγώ σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να μάθουμε ο ένας τι σκέφτεται ο άλλος ε, κάτι που βοηθά πολύ στις έρευνές μας. Αυτά, νομίζω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά όσοι μόλις ήρθατε στην αίθουσα. Συνιστώ να διαβάσετε την ετήσια έκθεση. Δεν είναι μόνο ένα ευχάριστο, μάλλον δεν είναι μόνο ένα χρήσιμο, αλλά και ένα ευχάριστο ανάγνωσμα. Ε, είναι, έχει κάποια χιουμοριστικά αποσπάσματα, σύνδεσμους με σχόλια Twitter κτλ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. So, so welcome colleagues. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε. Έχουμε τώρα την ώρα ψηφοφορίας. Παρακαλώ να τοποθετήσετε την κάρτα σας στο μηχάνημα. Οι ψηφοφορίες είχαν προγραμματιστεί για τις 4 και 20. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν ακριβώς την ώρα που προβλεπόταν. Διακόπτουμε για μερικά λεπτά. So it was nice to have. Ωραίο ήταν το διαλυματάκι μας. Ελπίζω να είστε έτοιμοι τώρα για να περάσουμε στην ψηφοφορία. Νομοδότηση λοιπόν σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών Μπεατρίθ Μπεθέρα η συγγήτρια 93 τροπολογίες κατατέθηκαν 10 συμβεβαστικές συνολικά για 76 τροπολογίες. Εκεί, μάλλον ο κύριος Χάναν θα κάνω μια δήλωση πριν περάσουμε στην ψηφοφορία. Μου έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να πω απλά ότι εκτιμώ το γεγονός ότι η σύγχυση μεταξύ αυτού του θύματος και της ευρωπαϊκής ε, ταυτότητας ε, ελήφθη και έτσι μπορώ να στηρίξω, όπως και όλοι φαντάζομαι, αυτή την έκθεση πλέον. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν τώρα στην ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία 1 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 78. Α, μάλιστα, όχι. Καταπέπτουν. Τροσυμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 34 ψήφι υπέρ, κατά, Α, υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει το λόγο για την προφορική αυτή τροπολογία. Όχι. Καλώς. Ψηφίζουμε λοιπόν. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω αλλά καλύτερα να ελέγξουμε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 49. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Υπάρχει προφορική τροπολογία. Όπως το βλέπετε και γραπτός. Θέλετε το λόγο. Υπάρχει πρόβλημα με τον ορισμό του European Legal Status, Ευρωπαϊκό Οικονομικό Καθεστώς. Γι' αυτό και είμαι κατά αυτής της προφορικής τροπολογίας και ζητώ να ψηφίσουμε την αρχική τροπολογία 49. Είναι κάποιος αντίθετος, λέει πρόεδρος, σε αυτή την προφορική τροπολογία. Amendment in favor. Ψήφι υπέρ της προφορικής τροπολογίας. Μάλλον του αρχικού, λέει πρόεδρος τώρα. Λοιπόν, εμπερδεύτηκα λέει η πρόεδρος. Ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο. Γιατί αυτό έχει γίνει δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική. Όχι. Τροπολογία 56. Όχι. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 70. Περιλαμβάνει προφορική τροπολογία. Υπάρχει κάποιος που θέλει το λόγο για την προφορική αυτή τροπολογία ή σας ικανοποιεί η γραπτή διατύπωση. Φαίνεται πως ναι. Ψηφίζουμε λοιπόν την προφορική τροπολογία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα λοιπόν περνάμε στην 53 τροπολογία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Το 54 ψήφι υπέρ κατά αποχές νομίζω απορρίπτεται να ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία για το 54 πέρας εγκρίθηκε αλλά ήταν αμφίροπτο αποτέλεσμα τροπολογία 60 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 77 υπέρ, κατά, αποχές, πρέπει να ελέγξουμε και την 77. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Καταπίπτει 84. Πηγαίνουμε λοιπόν στην 85 υπέρ. Κατά. Ποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 92. Σε δύο τμήματα σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα καταπίπτει, πάει αυτό. Πάμε στο δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο της σχέδιου Ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Δύο παραπάνω από το ΕΛΚ. Δύο. Τώρα ένας παραπάνω. Τώρα είμαστε εντάξει. Στις ψηφοφορίες κάποιος λέει το ίδιο συνέβαινε. Όχι. Λοιπόν, πέρασε της ψηφοφορίας. Και να συγχαρούμε την εισηγήτρια. Ομόφωνα εγκρίθηκε η γνωμοδότηση. Κυρία Μπεθέρη, θέλετε το λόγο, ορίστε παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην κατάρτιση αυτής της γνωμοδότησης. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά συνεντικό το όλο εγχείρημα, αναστήσαμε κοινέ θέσεις, δεν μπορούσε να γίνει άλλο διαφορετικά όταν μιλάμε για την ε, πρωτοβουλία για των Ευρωπαίων πολιτών. Ήταν πάρα πολύ ε, ελπιδοφόρο το αποτέλεσμα γιατί πιστεύω ότι έτσι μπορούμε να δώσουμε και τη σωστή απάντηση και ανταπόκριση στις ανησυχίες των πολιτών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερα τη Γραμματεία για τη δουλειά που έκανε, που ήταν πάρα πολύ σημαντική για να καταλήξουμε στις συμφωνίες. Γιουλιάνα, σε ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τη γραμματεία, την τόσο καλή γραμματεία που έχουμε. Και τώρα να περάσουμε στο υπαριθμό 19 σημείο. Πρέπει να αναβάλουμε το σημείο αυτό, διότι αποφάσισαν γι' αυτό οι συντονιστές να μην προχωρήσουμε, διότι υπάρχει ακόμη κάποια σύγχυση. Πρέπει να σεβαστούμε την προθεσμία για την προφορική τροπολογία, η οποία έχει οριστεί ε, στις 30 Ιουνίου, ε, Τρίτη, απόγευμα. Αναβάλουμε λοιπόν την εξέταση του θέματο αυτού, του σημείου αυτού και περνάμε στο επόμενο. Αναφορά επαριθμών 0944 2004 τη Σίλα Έλλης Βρετανικής Ιθαγένεια, για ε, ε εκ μέρου τη οργάνωση κάτι και κατά τοξικού χώρα που τα αφήσει αποβλήτων σχετικά με την προτιθέμενη αδυναμία του ΗΠΑ εφαρμόζοντα την οδηγία, τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων. <clears throat> Η αναφέρουσα είναι εδώ, η κυρία Έλλη, και στρέφομαι σε εσά για να σα δώσω το λόγο για την παρουσίασή σα. Το πολύ πέντε λεπτά. Συνάδελφοι, παρακαλώ προσοχή και σεβασμό προς την αναφέρουσα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αίθουσα και θέλω να της δώσω το λόγο. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Και για μένα και για τον Colin Wakefield που είναι πρόεδρο ε, της Πρωτοβουλία των Πολιτών ε, κατά του ε, ταφή, ταφής που έχει αποβεί τοξικός για την πόλη του Χότον Λεσπρίνγκ στην Αγγλία. Είναι μεγάλη μας χαρά που ερχόμαστε εδώ ξανά. Τα τελευταία 11 χρόνια, ε, από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, και έγινε καταγγελία στην Κομισιόν, έχουμε καταφέρει να δώσουμε 17 ατόμους από ε, στοιχεία τα οποία υποστηρίζουν την, ε, το αίτημά μας. Ότι δηλαδή οι πολίτες της Ευρώπης έχουν, είναι σε μειονεκτική θέση λόγω της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Έχει περάσει πολύ καιρό από το 2004. Επαναλαμβάνω ότι οι αρχέ του Ηνωμένου Βασιλείου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Σάντριλαντ και το ε, Γραφείο Περιβάλλοντο του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν αφήσει ε, να μολυνθούν οι ταμιευτήρε μια μικρή χώρα από την BIFA Waste Services, ε, που είναι η εταιρεία που διοικεί το χώρο υγειονομική ταφή παρά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τους χώρους υγειονομικής σταθής και την προστασία του περιβάλλοντος ε, ε, που έχει μεταφερθεί στο αγγλικό δίκαιο. Παρά τις διώξεις ε, που έκανε το Γραφείο Περιβάλλοντος για την μόλυνση και παρόμοιες λιγότερο θαραλές προσπάθειες από τις υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας υπήρξε ένα θάνατος παιδιού που θα μπορούσαμε να αποφύγει και ε, συνεχώς οι αρχές δεν καταφέρνουν να προστατέψουν τους πολίτες. Κάθε μέρα λοιπόν ε, μολύνονται μολύνεται το υδροφόρο ορίζοντα ε, και τα αποθέματα νερού που έχουμε λόγω αυτού του χίτα. Ο σταθμός του Stony Wait που χρησιμοποιούσε νερό από αυτόν τον υδροφόρο ορίζοντα, από αυτόν τον ταμιευτήρα πλέον δεν μπορεί να το κάνει και όλοι οι ταμιευτήρε μα έχουν καταστραφεί. Στην τελευταία συνεδρία της, Επιστρο... της Επιτροπής σας μας υποσχεθήκατε ότι θα ξεκινήσουν ασφαλιστικά και μέτρα και ότι θα κλείσει ο ΧΙΤΑ. Ε, μάλιστα δόθηκε η εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει κάτι τέτοιο και γυρίσαμε σπίτι μας με χαρά, θεωρώντας ότι δικαιώθηκαν οι πολίτες. Παρ' όλα αυτά τίποτα δεν συνέβη και ο λόγος ήταν ότι ο αξιωματούχος της Επιτροπή αρνήθηκε να λάβει ασφαλιστικά μέτρα κατά του Ηνωμένου Βασιλείου. μήπω είναι σύμπτωση που ο άνθρωπος αυτός ήταν ανώτατος αξιωματούχο στο δημόσιο, την κυβέρνηση δηλαδή του Ηνωμένου Βασιλείου πριν αναλάβει αυτή τη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και δεν θέλει να προσβάλλει τους τα προηγούμενα αφεντικά του. Τι δημοκρατία έχουμε όταν οι ευρωβουλευτές που είναι άμεσα εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι πληρώνουν για το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν, στην ουσία παραγωνίζονται από έναν δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος θεωρεί ότι είναι το αφεντικό και όχι ο υπηρέτης. Αυτός ο συγκεκριμένος δημόσιος υπάλληλος μας είπε πέρυσι ότι ε, είχε άλλη μία έκθεση από το Ηνωμένο Βασίλειο που ισχυρίστηκε ότι αποδείκνει ότι δεν υπήρχε πλέον μόλυνση από τον Χίτα και ότι το είχε κλείσει αυτός ο χώρος υγειονομικής ε, ταφής. Αυτό δεν ισχύει. Έχουμε αποδείξει ε, και στο παρελθόν τα ψέματα των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου. Μάλιστα μας είπε ότι θα μας έστελνε αντίγραφο της ε, εκθέσης το 2015. Δεν πήραμε τίποτα. Ενώ εμείς τα τελευταία 11 χρόνια Θέλουμε συνεχώς αποδείξεις στην Κομισιόν και στην Επιτροπή σας που είναι ακριβής. Έχουμε αποδείξει το δίκαιο του αιτήματό μας, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Έχουμε αειδιάσει. Έχουμε έρθει σήμερα εδώ ως μια ίστατη προσπάθεια για να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας και τα δικαιώματα των πολιτών. Σας ευχαριστούμε και τώρα ο λόγος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εκπρόσωπό της, τον κύριο Πολ Σπάιτ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πράγματι χρόνια κρατεί αυτή η αναφορά και σίγουρα οι αναφέροντες πολλά υπέφεραν όλη αυτή τη χρονική περίοδο. Ωστόσο, όλα τα δεδομένα τα οποία λάβαμε από τις αρμόδιες αρχές, όλα τα στοιχεία που μας έστειλαν αποδεικνύουν ή δείχνουν τέλο πάντων ότι σήμερα η κατάσταση φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί. Κατανοώ ότι και η Επιτροπή Αναφορών έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων πρόσφατα συμφωνούμε με, με τους αναφέροντες ότι υπήρξαν τις λειτουργίες τα τελευταία χρόνια. Το Ηνωμένο Βασίλειο πάντως ε, προέβαινε πάντοτε στις ε, απαραίτητες ενέργειες για την ε, διόρθωση των δυσλειτουργιών. Στα τέλη λοιπόν του 2014 έκλεισε την πιλωτική έρευνα η Κομισιόν σε αυτό το χώρο ταφής απορριμμάτων αλλά ζητούμε συνεχώς κάποια στοιχεία, παρακολουθούμε την κατάσταση, οπότε εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία θα παρέμβουμε εκ νέου στις ε, Βρετανικές Αρχές. Σε ό,τι αφορά τώρα τους ισχυρισμούς για την ε, μη ε, σωστή μεταχείριση. Όπως ξέρετε, εμείς πολλές φορές ασχολούμαστε με τέτοια ζητήματα, είτε παράνομες χωματερές, είτε νόμιμε, όπω στην προκειμένη περίπτωση που λειτουργούν όμω. Και πρέπει να σα διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει τον ίδιο χειρισμό. Ε, ισότιμα αντιμετωπίζει όλα τα κράτη, είτε είναι η Σλοβακία, είτε είναι το Βασίλειο, είτε οποιοδήποτε άλλο κράτο μέλο. Τέλο, πρέπει να σα πω ότι πράγματι στι τελευταία συνεδρία τη Επιτροπή Αναφορών υπήρξε κάποια σύγχυση για τα επόμενα βήματα ενδεχομένω κτλ. Το ζήτημα των ασφαλιστικών μέτρων υπευλήθη αίτημα κατά κάποιο τρόπο από την Επιτροπή σας. Είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται εκτάκτως και σε πάρα πολύ έκτακτες περιστάσεις. Πολύ ελάχιστες φορές χρησιμοποιήθηκε τα τελευταία 30-40 χρόνια και δεν θεωρούμε ότι θα ήταν και το κατάλληλο ε, μέτρο στην προκειμένη περίπτωση. Τώρα, για τις εκθέσεις οι Βρετανικές αρχές νομίζω ότι θα έρχονταν σε επαφή με τους αναφέροντες, θα τους έδιναν αντίγραφο της έκθεσής τους και αν δεν απατώμε έχουν στείλει τώρα τα έγγραφα που έστειλαν στο Κοινοβουλίο, τέλος πάντων έχουν πει ότι θα τα στείλουν στους αναφέροντες και αν δεν τα έχουν λάβει θα τα λάβουν σύντομα οι αναφέροντες. Ευχαριστώ. Now let's open the floor to members. I think... Ποιος συνάδελφος θα ήθελε τώρα το λόγο, νομίζω ο κυρία Κέρτον Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους αναφέροντες που ήρθαν εδώ από τη Ανατολική Αγγλία που είναι και η δική μου περιφέρεια για να παρουσιάσουν εκ νέου αυτή την υπόθεση. Πρόκειται για μια αναφορά που αποτελεί παράδειγμα, πώς να το πω, ίσως αποτελεί κομμάτι μιας ε, σειράς αναφορών που απογοητεύει προστατεύονται οι πολίτες από το πόσο βραδία είναι η ανάληψη δράσης ότι ουσιαστικά δημιουργούνται ψευδές προσδοκίες, ψευδείς προσδοκίες, συγγνώμη, και το είδαμε και σήμερα το πρωί στην ακρόαση που μιλούσαμε για τη λειτουργία των επιτροπών αναφορών σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολλές φορές δημιουργούνται ε, ψευδείς προσδοκίες λόγω της ε, ε των ενεργειών που παραλαμβάνονται. Ε, αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα και ευτυχώς έχουμε και κάποια καλά παραδείγματα. Ε, διότι είναι κρίμα να προκύπτει αγανάκτηση και απογοήτευση στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι ζουν ε, σε πάρα πολύ απαράδεκτα επίπεδα ρήπανσης και υπό πολύ κακές συνθήκες στις περιφέρειές έτσι εκτός πρακτικών να είμαστε προσεκτικοί για το μέλλον. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προκειμένη υπόθεση και την κατάθεση στο Χότον, είναι απογοητευτικό το ότι παρά το ότι υποσχέθηκαν να δώσουν τις εκθέσεις που υποτίθεται ότι είχαν ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, δεν διαβιβάστηκαν από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου στους αναφέροντες Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα τις πήραν. Τέλος πάντων αυτή την πληροφορία πολύ πρόσφατα λάβαμε. Μεγάλη καθυστέρηση λοιπόν σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των αναφερόντων. Εμείς κάναμε λίγο τη δική μας έρευνα, το δικό μου γραφείο δηλαδή, και από την ενημέρωση που είχαμε από τον Οργανισμό Περιβάλλοντος ε, είναι πάρα πολύ ψηλά των επιτρεπόμενων ε, τα επίπεδα ε, της αμμονίας. Και έχουμε ε, στοιχεία για το καλοκαίρι ότι καλά ήταν τα επίπεδα, τόσο προς σωστή κατεύθυνση, επισήμως όμως δεν ακούσαμε κάτι από την από την συγκεκριμένη αρχή και θα πρέπει οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να μας αναφέρουν την κατάσταση Υπάρχουν στοιχεία σίγουρα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να μπουν σε μεγαλύτερο βάθος, αν θέλετε. Δεν είχαμε χρόνο να μελετήσουμε όλα τα στοιχεία, γιατί και εμείς προσφάτως τα λάβαμε. Και ένα άλλο που θέλω να πω. Με χαροποιεί το γεγονός ότι θα σας πω, έχει πρώτα απ' όλα πενταετή σύμβαση ε, ο ανάδοχος ε, από το 2013 στο 2018. Αλλά νομίζω το Δημοτικό Συμβούλιο δεν δίνει παραπάνω προθεσμία. Πρέπει να έχει καθαρίσει αυτός ο χώρος και να κλείσει αυτός ο ΧΙΤΑ. Όσοι λοιπόν ενέχονται, όσοι μετέχουν εταιρεία, ο Οργανισμός Περιβάλλοντος, ε, το Δημοτικό Συμβούλιο και όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν πλέον αυτή την προθεσμία του 18. Είναι η τελευταία η καταληκτική προθεσμία και πρέπει να τηρηθεί. Γιατί έχει κρατήσει πραγματικά πάρα πολύ και δεν έχουν πλέον ε, υπομονή οι κάτοικοι. Και κάτι τελευταίο. δεν είναι μόνο μια κριτική προς αρχές του Βασιλείου. Νομίζω ότι υπήρξε και πρόβλημα διαφάνειας και από πλευράς κομισιών στο διάλογο που είχε με τους αναφέροντες. Και ήδη από την αρχή της υποβολής αναφοράς το βλέπουμε. Τους παρέκαμπταν από την αρχή τους αναφέροντες. Το είπαμε. Το είπε και η Κομισιόν, ε, ο είπε ο ίδιος ότι ενθάρρυνε, τι ενθάρρυναν τις αρχές να στείλουν αυτά τα έγγραφα. Μα αυτές, αυτά τα έγγραφα έπρεπε να τα πάρουν πρώτοι αναφέροντες. Δεν έπρεπε να φτάσουν εδώ ή να αναγκαστεί η Κομισιόν να ζητάει από τις αρχές της Τρόμας Βασιλή να στέλνουν αυτά τα έγγραφα. Είναι ένα θέμα δημόσιας υγείας, ρήπανσης. Η κομισιο να γνωρίζει τα επίπεδα της ρήπανσης και πρέπει η τοπική κοινωνία να μπορεί να κινητοποιηθεί. Έπρεπε λοιπόν αμέσως να είχε ενημερωθεί και να μην έρχονται εδώ συνεχώς να ρωτούν και να ζητούν αυτές τις πληροφορίες. Αυτό πραγματικά δημιουργεί ακόμη και περισσότερη απογοήτευση και τους κάνει να μιλούν για έλλειψη διαφάνειας και για να προχωρήσουμε και να δημιουργήσουμε ή να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη γιατί αυτή η αναφορά, επαναλαμβάνω, κρατάει πολύ καιρό, πολλά χρόνια. Για να γίνουν αυτά λοιπόν, πρέπει να δοθεί ένα τέλος, το σωστό τέλος όμως, από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Και θα πρέπει να υπάρξει και διάλογος με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Να υπάρξει και σωστή συνέχεια και παρακολούθηση το θέμα. Και μετά μόνο να αποφασίσουμε εμείς να κλείσουμε την αναφορά. I haven't seen anybody else asking for the floor. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος που ζητά το λόγο. Να σας ξαναδώσω λοιπόν το λόγο, κυρία Έλλης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω απλώς ότι σε αυτή τη φάση είμαστε και απογοητευμένοι με την απάντηση του κ. Σπέιτ, ο οποίο ε, ισχυρίζεται ότι τα πράγματα έχουν σταθεροποιηθεί, ε, η πρόσβαση στο νερό επίση. Αυτό σημαίνει ότι ελέγχεται το επίπεδο ρήπανση ε, στο 120 από το επιθυμητό επίπεδο. Είναι αυτό σταθεροποίηση, είναι σταθεροποίηση σε υψηλό επίπεδο μόλυνση για το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να τονίσω ότι δεν έχουν ληφθεί από το κράτος τα απαραίτητα μέτρα ε, και δεν είχαμε αυτήν την τόσο πρόσφατη έκθεση. Καταλαβαίνω ότι θα έπρεπε να ενημερωθούμε την Παρασκευή το Σάββατο αυτή τη εβδομάδα, αλλά ήδη η καθυστέρηση είναι πολύ μεγάλη για να μπορέσουμε να σχολιάσουμε για την ενημέρωση που θα λάβουμε σε αυτήν την συνεδρίαση τη Επιτροπή σα και ε, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου μας έχουν κρατήσει στο σκοτάδι όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούν. Η Επιτροπή αυτή θεώρησε ότι είναι σκόπιμο να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα για αυτή την περίπτωση κατά των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, ήταν ε, μια απόφαση, μια ενέργεια που θεωρήθηκε σκόπιμη, δεν ήταν κάτι που κρεμούσε, αλλά απορρίφθηκε από την Επιτροπή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν ε, λάβαμε καμία ενημέρωση. Μας άφησαν τελείως το σκοτάδι. Ταυτόχρονα ο χώρος ταφής ε, λειτουργεί ακόμη. Έχουμε δει χώματα, έχουμε δει ε, και άλλα υλικά να εναποτίθενται. Η βασική επιφάνεια έχει απλώς καλυφθεί. Ένα πολύ μικρό μέρος του δεύτερου χώρου έχει καλυφθεί με πολυεθαλήνη υψηλή πυκνότητας αλλά αυτό για τα ε, προηγούμενα ε, ισχύει εδώ 8 χρόνια. Είναι τελείως περιττή η ενέργεια αυτή και από ό,τι ξέρω υπάρχει μόνο μία τριετία περιθώριο για τη λειτουργία αυτού του χώρου ταφής. Θα θέλαμε λοιπόν πραγματικά αυτός ο χώρος ταφής να πάψει να χρησιμοποιείται κατά τις εκτιμήσεις έχει 17 χρόνια χρήσης πίσω του και πιστεύουμε ότι οι αρχές θα προσπαθήσουν να συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν. Η εταιρεία μάλλον με την έγκριση των αρχών του ΕΒ. Βασιλείου. Να ολοκληρώσω λέγοντάς σας ότι πριν από λίγο καιρό ε, ένας οργανισμός ε, περιβάλλοντος και ένας υπάλληλός του μας ζήτησε να μην εμποδίσουμε τη λειτουργία του χώρου αυτού. Θεωρεί ότι είναι επικίνδυνη η ε, τάση που τηρούμε με πολύπλοκες νομικές επιπτώσεις και ενδεχομένω με οικονομικές συνέπειες. Όμως η φήμη του οργανισμού αυτού πλήγει σοβαρά λόγω αυτής της τοποθέτησης. Μα πραγματικά Πώ να αφήσουμε τη φήμη, την καλή φήμη του οργανισμού περιβάλλοντο του Ρωμανού Βασιλείου να πλήττεται ενώ συμβαίνουν όλα αυτά. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρο, και εγώ σα ευχαριστώ και εκ μέρου των μελών τη Επιτροπή να ζητήσω πραγματικά συγγνώμη ε, για την καθυστέρηση. Η αναφορά αυτή εξετάζεται επί 11 χρόνια. Καταλαβαίνω ότι υπήρξε πολύ πόνο, πολλή ταλαιπωρία, πολλή δυσφορία και θυμό και ε, δικαιολογημένα. Ε, έχετε κάθε λόγο να αισθάνεστε έτσι. Είναι πραγματικά μια δυσάρεστη κατάσταση, διότι από ό,τι μου λέγεται έχουν ε, δεχτεί πίεση πέραν του ορίου ανοχής ε, οι περισσότεροι ε, άνθρωποι που μπλέκονται στην όλη υπόθεση. Και από την άλλη θα τρασπάλουμε να σας δώσουμε φρούτες ελπίδες. Ελπίδες ότι θα μπορούσαμε να βρούμε μια βιώσιμη λύση. Μακάρι να μπορούσαμε. Αυτό που μπορούμε όμως να κάνουμε είναι να μελετήσουμε αυτό το σύνολο εγγράφων, το οποίο λάβαμε μόλις χθες στη γραμματεία στις 7 το απόγευμα. Και δεν είχαμε αρκετό χρόνο ούτε στον πρώτο της γραμματείας, ούτε μεταξύ των συναδέλφων για να μελετήσουμε αυτά τα έγγραφα. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποστείλουμε επιστολή στις τοπικές και εθνικές αρχές, επισημένοντας ότι μας απασχολεί το όλο θέμα, βρίσκεται εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων μας, εντός του πεδίου ενδιαφερόντων της Επιτροπής αυτής, διότι πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και την ε, αξιοπιστία μας και να ενθαρρύνουμε τις αρχές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα αλλά στην τελευταία φράση αυτού του εγγράφου τη διαβάζουμε. Εντό εισαγωγικών. Για οποιοδήποτε ενέργειες και δράσεις συζητούνται, δεν προβλέπεται κάτι επιπλέον μελλοντικά στο άμεσο μέλλον. Εφόσον κάτι προκύψει θα ενημερώσουμε την Επιτροπή όπως δει. Αυτή είναι η τελική πρόταση. Προτείνω στους συναδέλφους αυτό και να κάνουμε. Να γράψουμε αυτές τις δύο επιστολές προς τις τοπικές και τις εθνικές αρχές και να παραμένουμε σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη γραμματεία μας για το θέμα αυτό. Η γραμματεία, ε, ο υπεύθυνο στη γραμματεία θα φροντίσει να έχει ανοιχτή γραμμή με την Επιτροπή αφού αναλύσει το έγγραφο. Αυτό θα ήταν ε, αποδεκτό για σας. Έλλης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, θέλουμε να τηρούμε θα ενήμεροι. Πρόεδρος, βεβαίως και θα το κάνουμε λοιπόν. Εγώ θα υπογράψω την επιστολή μόλις λάβει την τελική της μορφή και μόλις ληφθεί η απαραίτητη δράση. Εν τω μεταξύ θα σας ενημερώνουμε διαρκώς για το τι συμβαίνει. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε εδώ. σα ευχαριστώ για την υπομονή σας με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Μην ε, ε, πάψετε να πιστεύετε στην Ευρώπη. Επόμενο σήμερα τη μερικής διάταξης. Αναφορά 254 το 2013. για, την, για το χώρο απόθεση τοξικών αποβλήτων. Πάδοβα, Ιταλία. Ο Φιλίππο Ζόντιο είναι εδώ, ο αναφέρον, και θα του δώσω το λόγο, παρακαλώ. Το κτίριο της πρώην CNC εκτείνεται σε μια επιφάνεια 13.000 τετραγωνικών μέτρων. Σε αυτό έχουν σωρευτεί από το 2002 στο 2005 52.000 τόνοι ε, ιδιαίτερως επικινδύνων αποβλήτων. Στην εξωτερική έκταση 67.000 τετραγωνικών μέτρων έχουν ταφεί ε, τυχαία 3.500 τόνοι ε, των ίδιων αποβλήτων, ένα υλικό το οποίο πολύ πρόσφατα ε, το ε, έχουμε εκτάψει. Η περιοχή του Βένετο το 2009 αφιέρωσε 200.000 ευρώ για να μελετήσει τη μόλυνση του ε, δάφους και των υδροφόρων οριζόντων, αλλά αυτό δεν αρκεί. Η ανακαίνιση του κτηρίου το 2014 με 260.000 από τα 500.000 ευρώ που είχε προβλέψει η περιφέρεια του Βένετο δεν είναι μια οριστική λύση. Η κάλυψη των ρογμών στους τείχους και στη στέγη έδειξε επιπλέον ότι είναι επισφαλής οι συνθήκες λειτουργίας του κτηρίου και με την καταιγίδα που χτύπησε την, ε, έπληξε την περιοχή στις 13 Οκτωβρίου του 2014. Η σώρευση των υλικών αυτών που φτάνουν τα 6 μέτρα ύψος πιέζουν τους εξωτερικούς τοίχους απειλώντας την ε, σταθερότητα και τις φέρουσες κολόνες του κτηρίου με ε, αποτελέσματα διαβροτικά. Το νερό που περνά από τις ρογμές στην οροφή ε, σχηματίζει εσωτερικά δηλητηριώδεις λακκούβες και ριάκια νερού όπου καταλήγουν τα εκραίοντα ύδατα. Από τα 200.000 ευρώ των 500.000 που έχει αφιερώσει η περιφέρεια του Βένετο προβλέπεται μόνο το 3% των 52.000 τόνων των ιδιαίτερως επικίνδυνων αποκλήτων να μεταφερθούν. Εν τω μεταξύ επιδεινώνεται κατάσταση λόγω του κινδύνου στον οποίο είναι εκτεθειμένος ο χώρος, διότι βρίσκεται σε μια περιοχή υψηλού υδρολογικού κινδύνου. Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί πλημμύρες και πολλές φορές φτάνουν ως τα απόβλητα. Θα μπορούσε να προκύψει μια τεράστια καταστροφή για το περιβάλλον στη γύρω περιοχή και για την αγροτική παραγωγή, αλλά και για τους ε, ε, διάβλους, τους υδάτινους ε, διάβλους της περιοχής, που φτάνουν ως την ε, ε θάλασσα της Βενετίας. Ε, επίσης έχει πληγεί από στροβίλους αέρα το τελευταίο διάστημα η όλη περιοχή και το 2007 είχαμε και μία πυρκαγιά που ελέγχθηκε την τελευταία στιγμή. Θα μπορούσε όμως να έχει τεράστιες, τεράστιες καταστροφικές συνέπειες. Ο κίνδυνο τη περιβαλλοντική καταστροφή, στην οποία είναι εκτεθειμένο ο χώρο τη ε, πρώην CNC, ε, αφορά και μια περιοχή με μεγάλα αστικά κέντρα και μεγάλη αξία, όπου καταλήγει ούτω ή άλλω ε, στην Ευγάνια Λεκάνη. Και βεβαίω είναι εγγεγραμμένη στην περιοχή του κοινοτικού ενδιαφέροντος, ΣΥΚ. Σε μία δεκαετία η, αρχέ, η κατάσταση δεν έχει αλλάξει και οι Ιταλικές αρχές δεν έχουν προβλέψει το κλείσιμο του χώρου αυτού παρά ε, τα 10 ε, εκατομμύρια ευρώ που χρειάζονται. Τον Δεκέμβριο του 2014 η περιφέρεια του Βένετο έχει αφιερώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ στην υποτιθέμενη μεταφορά μέρους των αποβλήτων. Όμως το ποσό έχει μπλοκαριστεί σε επίπεδο ε, Υπουργείου Περιβάλλοντος και δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία αυτή παρόλο που ο χώρος αυτός είναι δημοσίου ενδιαφέροντος. Ζητούμε λοιπόν από τις αρχές των Βρυξελών να ε, εγκαλέσουν τις Ιταλικές αρχές και να κληθούν αυτές να επιλύσουν το πρόβλημα ακόμη και με ευρωπαϊκά κονδύλια. Πρέπει σύντομα να ληφθούν μέτρα γιατί μπορεί να υπάρξουν ανυπολόγιστε συνέπειε για την υγεία των πολιτών εκτός από την ε, ε, υπέροχη περιοχή αυτή των ε, θερμών πηγών που βρίσκεται το κτίριο της πρώην TNT. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα να δώσω το λόγο στην Επιτροπή και τον την εκπρόσωπό της, την κυρία Μανταλένα Καπρούσο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον αναφέροντα που βρίσκεται σήμερα εδώ και έκανε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση με φωτογραφικό υλικό. Η αναφορά έφτασε στην Επιτροπή του 2013. Μεταξύ του 2013 και 2014 εξετάσαμε το θέμα με ιδιαίτερη προσοχή και ήρθαμε σε επαφή με τις Ιταλικές αρχές, οι οποίες ε, απήντησαν ικανοποιητικά. Βάσει των ε, πληροφοριών που λάβαμε από τις Ιταλικές αρχές και αφού ασκήθηκε έλεγχος και ανακάλυψαν οι Ιταλικές αρχές ότι ο χώρος αυτός περιέχει εγκαταλελειμμένα απόβλητα, έχει κινηθεί ποινική διαδικασία. Η εταιρεία έλαβε την εντολή να καθαρίσει τον χώρο και πιο συγκεκριμένα οι αρχές διέταξαν τη λήψη των εξής μέτρων. 500.000 ευρώ οικονομική εγγύηση από την πλευρά της εταιρείας, 200.000 ευρώ για τον καθαρισμό μόνο το 2009 και 500.000 το 2011. Επιπλέον, οι Ιταλικές αρχές ενημέρωσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι διαδικασίες καθαρισμού έχουν ήδη ξεκινήσει και σήμερα ακούμε από τον αναφέροντα ότι τα κονδύλια αυτά για τα οποία μάθαμε ότι έχουν ήδη αποδοθεί προς αυτό το σκοπό δεν φτάνουν για να καλύψουν το συνολικό κόστος καθαρισμού. Να θυμίσουμε στον αναφέροντα και στο Κοινοβούλιο ότι η Επιτροπή δεν έχει λάβει περαιτέρω πληροφορίε σε σχέση με την αναφορά αυτή από το 2013 και το 2014. Οπότε η δική μας έρευνα σε αυτή τη φάση έχει λήξει. Εάν ο αναφέρον έχει περαιτέρω πληροφορίες, μπορεί να μας τις προωθήσει και εμείς θα φροντίσουμε να τις μελετήσουμε και να προχωρήσουμε αναλόγως και ενδεχομένως με περαιτέρω έρευνα εφόσον χρειαστεί. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Εύη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση προφανώς σοβαρότατη. Αξίζει όλη μας την προσοχή. Διότι αν είναι αλήθεια Ακόμη μάλλον και να αληθεύει ότι δόθηκαν κάποιε εγγύσει για την επίλυση του προβλήματο, ταυτόχρονα ε, αληθεύει ότι η μαρτυρία που είχαμε σήμερα, το τι συμβαίνει δηλαδή σήμερα στην πράξη, θα πει ότι στην πραγματικότητα δεν έχει βρεθεί λύση. Είναι λοιπόν σημαντικό να παραμείνει ανοιχτή η εξέταση τη αναφορά αυτή για να έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία και τη βεβαιότητα που να μα επιτρέπει να πούμε ότι κάτι άρχισε να γίνεται για να βρεθεί μια λύση. Σήμερα αυτό δεν συμβαίνει να θυμίσουμε πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η περιοχή, περιοχή που απειλεί ολόκληρη έκταση, έκταση η οποία βασίζεται στη γεωργική παραγωγή, ε, παραδοσιακών προϊόντων, στην έλευση τουριστών λόγω των θερμών πηγών και είναι και ένα παραθυριστικό κέντρο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ονομάσουμε καρκίνωμα αυτό που συμβαίνει σε αυτό το χώρο, σε αυτό το πρώην εργοστάσιο ε, είναι σαφέ ότι πρέπει οι Ιταλικέ Αρχέ να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθούν την προστασία τη ευρύτερη έκταση και να καθαρίσουν αυτό το χώρο. Τα 500.000 ευρώ που έχουν ε, αφοσιωθεί στι ε, γεωτρήσει για να διαπιστωθεί η υγειονομική κατάσταση του χώρου δεν έχουν γίνει ακόμη. Δεν έχουν δαπανηθεί τα θέματα αυτά, τα κονδύλια αυτά. Άρα σίγουρα υπάρχει καθυστέρηση. Χρονοτριβούν οι αρχές. Οι γεωτρήσεις αυτές είναι απαραίτητες ε, και πρέπει να γίνουν στο δυνατόν συντομότερα. Οπότε ζητώ η εξετάσταση της αναφοράς αυτής να παραμείνει ανοιχτή. Πρόεδρος. Άλλος κανείς θέλει το λόγο. Η κυρία Σκαρντίνη. Γκαρντίνη, συγγνώμη. Και μετά η κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ. Και εγώ να ευχαριστήσω όσους ήρθαν εδώ για να υποβάλλουν στην κρίση της Επιτροπής Αναφορών ένα τόσο ε, ευαίσθητο θέμα. Νομίζω το να έχουμε πολίτες με ευαισθησίες, με τέτοιες ευαισθησίες που προστρέχουν ε, στα θεσμικά όργανα με σκοπό να προστατεύσουν ε, και να διασφαλίσουν το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, δείχνει ότι οι καιροί έχουν αλλάξει, έχουν βελτιωθεί. Ο πλανήτης μας σιγά σιγά θα βρίσκεται σε καλύτερα χέρια από ό,τι φαίνεται. Εγώ είμαι από την Πάντοβα, οπότε γνωρίζω καλά τις ε, περιοχές για τις οποίες μιλούμε. Είναι όντως περιοχές ε, με ιδιαίτερη αξία και από πλευρά υδρολογικής ε, με ιδιαίτερες ανάγκες. Πρέπει λοιπόν η προσοχή μας να είναι τεταμένη. Ε, και εγώ θα φροντίσω επιστρέφοντας αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ιταλία να συζητήσω το κατά πόσον ε, οι τελευταίες ανησυχητικές ειδήσει που ακούσαμε ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Διότι το μισό εκατομμύριο ευρώ που έχει προβλεφθεί ο Σκοντήλη δεν μου επιβεβαιώθηκε από τις περιφερειακές αρχές με τις οποίες μίλησα την περασμένη εβδομάδα. Ή είναι πρόσφατη απόφαση ή δεν είχε ληφθεί καν. Οπότε ε, ελπίζω αυτό να το διαλευκάνω σύντομα και να ισχύει αυτό που ακούσαμε σήμερα. Σε ό,τι αφορά τα όσα όντως μπόρεσα να εξακριβώσω, θα έτεινα να θεωρήσω ότι το θέμα βρίσκεται υπό έλεγχο πλέον, όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι πράγματι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές ε, παρακολουθούν από το 2005 την όλη κατάσταση και έχουν ε, προχωρήσει σε πολύ συγκεκριμένε δράσεις. Ε, πληροφορούμε ότι σήμερα ο χαρακτηρισμός, ο περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός της περιοχής είναι Μάλλον, είτε ε, ως προς το, τα χαρακτηριστικά των ε, περιβαλλοντικών στοιχείων ή τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων που έχουν ε, αποτεθεί εντός του στεγασμένου χώρου είναι σε καλή κατάσταση. Από το 2013 ο Δήμος της Περνούμια έχει αναλάβει την ευθύνη όλων των διαδικασιών εξυγίανσης και ο Όμιλος έχει επίσης αναλάβει την ανακαίνιση του στεγασμένου χώρου. Οπότε θεωρείται ότι οι κατεπίγουσες ανάγκες ε, εξαιτία της περίπτωσης ε, κατάρρευσης του χώρου έχουν ξεπεραστεί. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν βέβαια τα απαραίτητα κονδύλια για την ε, μεταφορά των αποβλήτων, αλλά δεν είναι 10-12 εκατομμύρια η ανάγκη. Ο μιλός με διαγωνισμό ε, που σκοπό έχουν να προχωρήσουν σε ε, εκταφή και μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων. Στο διαγωνισμό η τιμή που καθορίστηκε ήταν 90 ευρώ ένα τόνο ε, αποβλήτων. Δεν φτάνουμε λοιπόν σε ένα τελικό κόστος 10-12 εκατομμυρίων, αλλά 5 ή 7 εκατομμύρια ευρώ συνολικό κόστος. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να παραδεχτούμε το πόσο ευαίσθητο είναι το θέμα, αλλά αρκεί να πούμε στις αρχές ότι πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τη δέουσα προσοχή, τις εξελίξεις για να μην υπάρξουν επιπτώσεις στις συντροφόρες λεκάνες των γειτονικών δήμων και κοινοτήτων. Αυτό θα ήταν όντω ιδιαίτερο επικίνδυνο. Νομίζω όμω ότι οι αρχέ που είναι ήδη τόσο δραστήριε και έχουν προχωρήσει τόσο πολύ στην αντιμετώπιση του θέματο, απλώ πρέπει να λάβουν την έκκληση να εντείνουν τι προσπάθειέ του και ίσω και την απόδοση κονδυλίων τα οποία να αυξηθούν ενδεχομένως περαιτέρω με τις ανάλογες γραμμές του προπολογισμού εντός του λειτουργικού προγράμματος για την περιφέρεια από τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά σε αυτή τη φάση πρέπει να συνεχίσει ευανιστικά η παρακολούθηση. Η κατάσταση όμως σήμερα βρίσκεται υπό έλεγχο. Όπως ε, επιστρέφω στην πόλη μου το Σαββατοκύριακο θα φροντίσω να πληροφορηθώ ακριβώς τι συμβαίνει και προσωπικώς θα λάβω μερίμνα για να ε, ενημερωθώ για το όλο ζήτημα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Άουκεν. Απλώς ε, να πω ότι όντας εδώ και ακούγοντας ε, καταλαβαίνω ότι είναι λίγο περίεργο να είναι εκεί τα λεφτά και να μην φέρνουν ευτυχία και να μην συμβαίνει τίποτα μάλλον και μετά να ξανάρχονται χρήματα και πάλι να μην γίνεται τίποτα. Ελπίζουμε κάτι να συμβεί. Λέτε στη γραπτή σας απάντηση ότι και τώρα πάλι μας είπαν ότι θα κάνουν κάτι. Και αυτό ακούγεται καλό. Ο τρόπος ε, που αντιμετωπίστηκε η διαχείριση των αποβλήτων στην Ιταλία τα τελευταία χρόνια, να το πούμε έτσι, πραγματικά είναι λίγο περίεργο, αλλά ελπίζω κάτι να συμβεί. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να παρακολουθούμε τι συμβαίνει. Όλο και περισσότερα χρήματα δίνονται χωρίς να ρωτάμε τι έγινε με τα προηγούμενα χρήματα. Με την προηγούμενη πρωτοβουλία. Μόνο και μόνο επειδή μας λένε ότι θα κάνουν κάτι. Ας το παρακολουθούμε λοιπόν και είναι καλό που τουλάχιστον όλο και περισσότεροι λένε ότι κάτι θα γίνει. Μίστη Βαλέσσα. Ο κύριος Βαλέσα. Ήταν μια μεγάλη μέρα. Προσπαθώ να καταλάβω. Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι αρμόδιες Ιταλικές αρχές έκαναν τις κατάλληλες ε, δράσεις ώστε να καθαριστεί η περιοχή και δόθηκαν και χρήματα για την απορρίπανση. Και καταλαβαίνω από την Κομισιόν ότι λόγω της δράσης των αρχών έχει κλείσει η έρευνα της Κομισιόν. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εμείς ως Επιτροπή αναφορών. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις και αυτό λένε και οι εκπρόσωποι της Κομισιόν. Αν όμως ο Ετών έχει κάποια στοιχεία καινούρια που μπορούν να ξανανοίξουν την έρευνα διότι έχει κλείσει η έρευνα από την Κομισιόν, έχω το εξή ερώτημα. Μπορούμε να αφήσουμε ανοιχτό το αίτημα, αλλά αν έχει κλείσει η έρευνα της Κομισιόν, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε ως Επιτροπή. Από τη στιγμή που έκλεισε λοιπόν ε, η Κομισιόν την υπόθεση, πρέπει και εμείς να κλείσουμε την αναφορά, θεωρώ κι εγώ. Εκτός αν υπάρχουν νέες ε, εξελίξεις ή μάθουμε κάτι άλλο που μας λέει ότι πρέπει να ξανανοίξουμε. Κυρία Σκαρδίνη. Γκαρντίνη, ευχαριστώ. Να προσθέσω απλώς κάτι, διότι είναι περίεργο να μιλούμε για ένα γεγονός μια υπόθεση που αφορά μια χώρα για μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο χώρο εναπόθεσης τελικά ε, δακτυλοδεικτείται μια ολόκληρη χώρα. Είναι πολύ άδικο αυτό. Έχουμε και άλλες περιοχές με προβλήματα και δυσκολίες, αλλά αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Η δική μου όμως η περιοχή, η δική μου περιφέρεια έχει αριστεία. Είναι ε, σε μια από τι πρώτε θέσει για τη διαχείριση αποβλήτων και ξεπερνά πολλέ άλλε χώρε τη Ευρώπη. Η ανακύκλωση με την αποκομιδή των ε, βιοδιασπόμενων, των υγρών, των ε, ε, πλαστικών και ούτω καθεξής στην περιοχή μου είναι από τι καλύτερες στην Ευρώπη. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να φύγεται η τιμή μια ολόκληρη χώρα μέσα από μια συγκεκριμένη περίπτωση. Ευχαριστώ. Ναι, ζητώ συγγνώμη. Η δική μου πρόθεση δεν ήταν να προσβάλλω κάποιον. Ξέρω ότι υπάρχουν περιοχές στην Ιταλία που ε, πραγματικά γίνεται καλή διαχείριση των αποβλήτων. Όχι μόνο στην Καμπανία, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη όμως μας λένε ότι τα πράγματα είναι καλά, αλλά όταν πάμε εκεί είναι καταστροφή. Βλέπεις τους πολίτες τους μιλάς και πραγματικά κατανοείς ότι κανένας δεν είναι ικανοποιημένο. Χαίρομαι που ακούω ότι υπάρχουν καλά μέρη. Δεν θα έπρεπε να το πω έτσι, τέλος πάντων δεν είχα πρόθεση να σας προσβάλλω. Maybe you two can go out and have a... Μήπως οι δυο σας να βγείτε και να πιείτε ένα καφεδάκι. With absolutely Μόνο ζάχαρη, χωρίς καθόλου δηλητήριο. Δεν βλέπω άλλους ε, συναδέλφους να θέλουν να μιλήσουν. Έχω αυτή την πρόταση που λέει να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά και υπάρχει και μία πρόταση να την κλείσουμε. Εφόσον οι υπηρεσίες της Κομισιόν αποφάσισαν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα και δεν θέλουν να ερευνήσουν περαιτέρω την υπόθεση. Αυτό μας είπε η γραμματεία της Κομισιόν της Προάλλες. Μπορούμε να κάνουμε το εξής. Εμείς ως Επιτροπή Αναφορών να στείλουμε και πάλι μια επιστολή στις Ιταλικές Αρχές όπου θα καταγράφουμε την κατάσταση και θα αναφέρουμε αυτά που είπε ο αναφέρον. Επίσης, να αναφερθούμε στην αλληλογραφία που υπάρχει και να πούμε ότι παρακολουθούμε το τι συμβαίνει, αλλά δεν μπορούμε να κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή, καθώς δεν υπάρχει επί της ουσίας κάτι νέο σε αυτή την υπόθεση. Να το κάνουμε αυτό και μετά να κλείσουμε την αναφορά. Κυρία Ειδη, τι λέτε. Νομίζω ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η εξέταση της αναφοράς αυτής μέχρι να λάβουμε απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να έχουμε τα στοιχεία για να δούμε πώς προχωράει η διαδικασία υλοποίησης. Μόνο τότε θα μπορούμε να την κλείσουμε. Και υπέρ και κάτι ακόμη. Δεν μπορούμε να λάβουμε απόφαση, διότι λείπουν και άλλες ομάδες. Και το να κλείσουμε την εξέταση της ε, αναφοράς χωρίς την γνώμη άλλων ομάδων μου φαίνεται άδικο. Χωρίς την παρουσία άλλων λοιπόν θα ήταν σοβαρή απόφαση και δεν θα ήθελα να έχουμε ένα τέτοιο σοβαρό κίνδυνο για ρήπανση από απόβλητα χωρίς να είναι σαφές ότι πρέπει να κλείσει όλη η διαδικασία. Θα ήθελα λοιπόν να περιμένουμε. Κυρία Βαλίνα. Ευχαριστώ. Συμφωνώ να αποστείλουμε την επιστολή και να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά μέχρι ότου αρχίσει να λύνεται το πρόβλημα. Όλοι γνωρίζουμε πώς ε, λειτουργούν τα πράγματα, άρα Καλύτερα να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά, να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μπορούμε να κλείσουμε την αναφορά. Κύριε Άουκεν, επίσης νομίζω ότι το συμπέρασμα εδώ είναι να μην μείνει ανοιχτή αναφορά γιατί στέλνουμε και ένα μήνυμα ότι παρακολουθούμε την κατάσταση. Πολλές ε, αναφορές κλείνουν όταν ε, πλέον έχουμε παρακολουθήσει ότι η κατάσταση είναι ε, ότι η δικασία έχει ολοκληρωθεί. Εμείς όμως θέλουμε να διαπιστώσουμε ότι δεν μας έχουν πει μόνο λόγια του αέρα. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουν ότι παρακολουθούμε την κατάσταση και ελπίζουμε να μπορέσουμε να κλείσουμε την αναφορά μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, αλλά είναι πολύ καλύτερο να παραμείνει προς το παρόν ανοιχτή η ανάφορα. Και δεν ξέρω ποιο επιχείρημα θα μπορούσε να μας πείσει να την κλείσουμε την αναφορά τώρα. Okay, let's do the following. Ωραία, άρα παραμένει ανοιχτή η αναφορά για να παρακολουθούμε τη διαδικασία καθαρισμού για την οποία μας ενημερώνουν. Στέλνουμε επιστολή στις αρμόδιες αρχές της Ιταλίας για να αναφερθούμε και στο διάλογο την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε σήμερα στην Επιτροπή μας. Προσπάθησα να ακούσω τις διάφορες προτάσεις. Δεν μπορούμε να κλείσουμε την αναφορά, όμως ορισμένοι από εσάς είστε συντονιστοί. Ποιο είναι το μάθημα για εσάς να φροντίσετε στην Επιτροπή σας να έρχονται τα μέλη από τις ομάδες σας. Είναι απαράδεκτο να μην εκπροσωπούνται ε, διάφορες ομάδες. Το ΕΛΚ ε, είναι εδώ, η Πράσινη εδώ, αλλά η δική μου ομάδα δεν είναι εδώ για παράδειγμα. Λείπουν οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες. Α, έχουμε ένα μέλη, όχι το συντονιστή όμως. Τέλος πάντων. Είναι μια μεγάλη επιτροπή αυτή δεν μπορεί κανεί από εσά να δικαιολογήσει ότι είναι 5-6 μόνο εδώ παρόντε από όλα τα μέλη που είναι γεγραμμένα στην Επιτροπή. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε του συναδέλφου μα να συμμετέχουν στι εργασίε τη Επιτροπής μα πολύ περισσότερο, πολύ πιο ουσιαστικά. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε με το σημείο αυτό και περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσιας διάταξης. Έχουμε λοιπόν την αναφορά 921 του 2012 για τη μη μεταφορά στην ειδική νομοθεσία της οδηγίας σχετικά με τον οργάνωση του χρόνου εργασίας. Ρουμανία. Δεν είναι παρόν να αναφέρον, δίνω το λόγο στον, στην Σάσα Γκάρμπαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2011 η Κομισιόν έλαβε καταγγελία από τον αναφέρον ότι τα δικαιώματα ετήσιας άδειας των υπαλλήλων στην Διεύθυνση για την Προστασία των Παιδιών στην Ρουμανία είχαν μειωθεί, μειωνόταν κατά μία μέρα για κάθε δέκα μέρες άδειας ε, ασθένειας. Αυτό φυσικά δεν συνάδει με το άρθρο 7 της ε, ε, οδηγίας για το χρόνο εργασίας που μιλάει για ένα ελάχιστο αιτήσιας άδεια, ειδικότερα στο ε, θυμικό δίκαιο της ε, περίπτωση της υπόθεσης Σούλτ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αναφέρεται ότι πρέπει οι άνθρωποι αυτοί στην ουσία να παίρνουν αιτήσια άδεια όταν ας πούμε έχουν ασθενήσει και αν μία περίπτωση ε, ασθένειας συμπέσει με την άδεια ε, διακοπών, τότε δεν χάνει την άδεια διακοπών. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή ήρθε σε διαβούλευση με τις Εθνικές Αρχές το 2013 για να μπορέσει να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα για το ε, νομικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο και από εκεί στην ουσία είδαμε ότι στον εργατικό κώδικα, στο άρθρο 451 ε, του Ρουμαν... της Ρουμανίας, ε, ήταν προβληματικό γιατί λέει ότι η ετήσια άδεια διακοπών είναι αναλογική με τη δουλειά που κάνεις. Δηλαδή, αν ασθενήσεις, δεν έχεις ετήσια άδεια. Και ε, φαίνεται ότι Υπήρξαν και κάποια κυβερνητικά εντάλματα που όριζαν το τι θα γίνει με το χρόνο εργασίας ανθρώπων που δεν συμμορφώθηκαν με το άρθρο αυτό της οδηγίας και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Έκλεισε λοιπόν η Κομισιόν την ανταλλαγή πληροφοριών σε πιλωτικό επίπεδο που είχε με τη Ρουμανία και έστειλε μια επίσημη επιστολή προειδοποίησης πέρυσι τον Φλεβάρη. Είναι το πρώτο στάδιο στη διαδικασία παραβίασης, όπως γνωρίζετε. Οι ε, ρωμανικές αρχές απάντησαν ενημερώνοντας την Κομισιόν ότι δεν αμφισβητούσαν την ανάλυση. Όντως είπαν και αυτές ότι υπήρχε ασυμβατότητα και ότι θα αλλάξει το νομικό πλαίσιο. Τώρα λοιπόν φέτος το Γενάρη άλλαξε ο εργατικός κώδικας και τώρα λέει συγκεκριμένα ότι οι περίοδοι προσωρινής ε, αδυναμίας εργασίας ε, θεωρούνται περίοδοι δραστηριότητας, οπότε συνεχίζεις να ε, έχεις αιτήσει άδεια εργασίας για αυτές τις ημέρες. Επίσης, αν έχεις άδεια ασθένεια, η οποία συμπέσει με την άδεια διακοπών, τότε μπορείς να αλλάξεις ε, την ετήσια άδειά σου και αν παραμείνεις ασθενής για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, σωρεύεις τις ημέρες της ετήσιας άδεια που μπορούν να πάνε παραπέρα και για 18 ολόκληρους μήνες, παραπάνω από ό,τι στην ουσία ορίζεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Άρα αυτό είναι ένα καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι εθνικές αρχές επίσης μας ενημέρωσαν ότι τώρα θέλουν να τροποποιήσουν και τα κυβερνητικά διατάγματα και ότι και από ό,τι φαίνεται αυτό το μήνα κατέθεσαν ένα προσχέδιο το οποίο θα εγκριθεί μέχρι τα τέλη του έτους και οι υπηρεσίε της Κομισιόν θυμίζουν στις εθνικές αρχές ότι οι κυβερνητικές αποφάσεις πρέπει και αυτές να αλλάξουν για να μπορέσουν να συνάδουν με τις αλλαγές στον εργατικό κώδικα. Θα κλείσει η διαδικασία παραβίασης από την Κομισιόν μόλις έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την ε, συμφωνία νομοθεσία ε, και όλων αυτών των στοιχείων που την απαρτίζουν στη Ρουμανία με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αλλά να πω ότι έχουν γίνει τα σωστά βήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε την επιστολή επίσης εδώ του αναφέροντος του κυρίου Σόριν Στέλιαν Τόροπ ο οποίος λέει ότι λυπάται πολύ που δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ. Είναι μια αναφορά αυτή για την οποία θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, όχι τελείως, αλλά για το αποτέλεσμα. Προτείνω λοιπόν να κλείσουμε αυτή την αναφορά και να το κάνουμε βάσει του γεγονότος ότι είναι μια success story της Επιτροπής μας. Ο αναφέρον έδωσε το θέμα το 2012. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε ε, αναφέροντας και διαπιστώνοντας ε, την ε, παραβίαση ως προς την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδη... αντίστοιχης οδηγίας έστειλε μια επίσημη επιστολή προειδοποίησης η οποία είχε ως αποτέλεσμα να διορθωθεί το πρόβλημα και έκλεισε το ζήτημα από τη δική μας πλευρά. Μπορούμε να στείλουμε το φάκελο στην Επιτροπή Απασχόλησης με τα δικαιολογητικά αλλά και στην αντιπροσωπεία, την αντιπροσωπεία της Ρουμανίας ζητώντας τους ευγενικά να παρακολουθήσουν αυτό το ζήτημα. Αυτό λοιπόν είναι ένα απλό ζήτημα, είναι η τελευταία μας αναφορά για σήμερα. Δεν συμφωνείτε κύριε Πιτέρα. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Γιατί θα έλεγα να κλείσουμε την εξέταση της αναφοράς αυτής. Τον Δεκέμβριο το Κοινοβούλιο της Ρουμανίας ενέκρινε νέο εργασιακό κώδικα, ο οποίος άρχισε να ισχύει ήδη και το πρόβλημα αφαίρεση σήμερα από την ετήσια άδεια έχει επιληθεί άλλα προβλήματα επίσης, οπότε χάρη στον εργατικό, εργασιακό κώδικα αυτά είναι ε, πλέον παρελθόν. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Στην επιστολή του αναφέροντος βλέπετε ότι έχουμε έναν αναφέροντα ε, που είναι επιτετέλους ικανοποιημένο. Δηλώνει ότι εάν η Ρουμανία δεν ήταν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί το πρόβλημά του να έχει παραμείνει άλυτο ή αναπήλυτο. Αλλά θέλει να ευχαριστήσει τους ευρωπαϊκούς ε, θεσμούς που εξυπηρέτησαν την ε, εξέφραση λύσης. Πολύ κομψό εκ μέρους του, αλλά εξέφρασε και τη λύπη του, διότι χρειάστηκε τόσο πολύ καιρός για να επιληθεί αυτό, μια τριετία. Στην Επιτροπή μας όμως πρέπει να σημειώσουμε και τα παράπονα και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, έχουμε ήδη προχωρήσει πιο γρήγορα, είμαστε πιο ε, στην εξέταση των αναφορών, έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά ε, συνάδελφοι, ε, έχουμε κουραστεί βέβαια από το πρωί, αλλά είμαστε πάλι σε καλή διάθεση. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους και πολύ εγκαίρως μπορούμε να κλείσουμε, εκτός αν θέλει το λόγο κάποιος, ο Ευχαριστώ τίποτα σημαντικό, απλώ να κλείσουμε την εξέταση τη αναφορά, θέλω και εγώ να πω. Και αν δείτε την αίθουσα, έχουμε ακόμα λιγότερου βουλευτέ από ότι ε, στι προηγούμενε αναφορέ. Κάποιο είπε ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε την ε, εξέταση τη αναφορά γιατί είμαστε τόσοι λίγοι. Τέλος πάντων, απλώς για να το παρατηρήσω, μια πολιτική παρατήρηση ήταν. Ναι, ήταν, είναι όμως πολύ ξεκάθαρη η περίπτωση αυτή, ενώ ε, οι άλλοι δεν ήταν. Η πρόταση ίσως αμφισβητήθηκε από πολλούς, απλώς δεν ήταν αρκετή ώστε να το πράξουν. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συνεδρία και θα σας δω την επόμενη φορά.